Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εγώ φταίω. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου και ορισμός συγητών. Δεν θα χρειαστούν πολύ χρόνο γιατί δεν υπάρχει κανείς βέβαια να ορίσουμε. Όσον αφορά λοιπόν τον ε, ορισμό αιωνσίτων, έχουμε δύο συμφωνίες ε, για τις αεροπορικές μεταφορών με το Μακάο και τη Σρι Λάνκα και η απόφαση των συντονιστών είναι ο πρόεδρος να ασχοληθεί με αυτά. Μετά είχαμε κάποιες γνωμοδοτήσεις που συζητήσαμε. Η απόφαση των συντονιστών ήταν να μην γίνει καμία ενέργεια. Το ένα ήταν έγγραφο εργασίας για την ενιαία αγορά, το άλλο η ανακοίνωση για την ε, προσαρμογή της πολιτικής ε, εμπορίου και επενδύσεων για τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ε, απλοποίηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Επιτροπή Προϋπολογισμού, οπότε είπαμε καμία ενέργεια. Επίσης, ε, επικοινωνίες και η θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, οπότε ούτε και εκεί πέρα θα κάνουμε κάποια ενέργεια όσον αφορά τις μελέτες. Οι συντονιστές ε, συμφώνησαν ε, να κάνουμε πέντε μελέτες η μία για το καμποτάζ το οδικό, η άλλη για τον αντίκτυπο των βιοκαυσίμων, κοινωνικές συνθήκες στις οδικές ε, μεταφορές, μεγάλα έργα τέντη και βιομηχανική κληρονομιά, τουρισμός για αγροτικές περιοχές. Αλλά συμφωνήσαμε πως εάν η ΣΤΟΑ αναλάβουν μία από αυτές τις μελέτες, ειδικά για τα βιοκαύσιμα, θα απελευθερωθεί μία άλλη μελέτη για μας. Συγγνώμη, κυρία. Αγροκαύσιμα τα λέμε τώρα. Α, συγγνώμη. Α, γιατί να μην λέμε τη λέξη βίο που είναι καλή. Αγροβιοκαύσιμα μάλιστα. Η μπορεί να μας πει και να έχουμε εμείς μια άλλη έκθεση. το δελτίο των διακαυσίμων, το δελτίο, με συγχωρείτε, της ε, επιτροπολογίας, για τις ε, ακροάσεις ε, αποφασίσαμε να γίνει μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Βιομηχανίας για το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη το πρωί της 24ης Απριλίου και επίσης θα εξετάσουμε το θέμα της ε, ακρόασης 3η 8 Μαΐου το πρωί για τις κατευθυντήριες γραμμές διευρωπαϊκών δικτύων και το απόγευμα για το πακέτο των αεροδρομίων. Πρέπει ακόμα να βρούμε ποια θα είναι η αίθουσα, αλλά θέλουμε 8 Μαΐου να έχουμε ακρόαση το πρωί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το απόγευμα για τα αεροδρόμια. Επίσης, ο κύριος Μπρίνκχορστ, ο συντονιστής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ε, απέστειλε μία επιστολή ως αποτέλεσμα ενός ε, ε, αιτήματος κατοίκων μιας περιοχής μιας αναφοράς των κατοίκων. Ναι, θα τα τελειώσω και μετά. Λοιπόν, οι συντονιστές ε, που είχαν ερωτήσεις ε, για την επιστολή του κυρίου Μπρινκχόρστ μπορούν να τις ε, απευθύνουν σε μένα και εγώ θα προωθήσω τις ερωτήσεις στον κύριο Μπρινκχόρστ. Και επειδή βεβαίως η αναφορά είναι απευθύνεται στο Κοινοβούλιο, πρέπει να πάει στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών για να γίνουν τα δέοντα. Και μετά βεβαίως ε, θα πούμε τα λοιπά στον κύριο Μπρινκχόρστ. Οι συντονιστές συμφωνούν η κυρία Τσίκαο να παραμείνει η αρμόδια για την ενσωμάτωση πολιτικής ε, των ε, φίλων. Στα διάφορα συζητήσαμε όντως διάφορα πράγματα και πολλά για την διασυνοριακή εφαρμογή ζήτησαν οι συντονιστές ο πρόεδρος να απευθύνει επιστολή στον κύριο Κάλλας για να ξεκαθαρίσει νομική βάση για την οδηγία αυτή. Για την κινητικότητα, την εβδομάδα κινητικότητας ε, αποφασίσαμε να τιμήσουμε την εβδομάδα αυτή 16 με 22 Σεπτεμβρίου με το να συμπεριλάβουμε μια παρουσίαση για την ε, κινητικότητα και την αστική κινητικότητα στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου και πάλι οι συντονιστές ζήτησαν να απευθύνω μία επιστολή στον πρόεδρο Σούλτς για να παίξει το κοινοβούλιο πιο ενεργό ρόλο στην εκδήλωση αυτή. Γιατί στο κυρία Τσικάου και ο κύριος Κάντσιαν που μας εκπροσωπούν θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις στους συντονιστές για έγκριση στην ε, συνεδρίαση του Μαρτίου μετά για τα μεγάλα φορτηγά, τα γιγαντιαία φορτηγά μου ζητήθηκε να έρθω σε επαφή με τον κύριο Κάλλας για να εκφράσουμε την ανησυχία μας για αυτά τα οποία ακούγεται ε, ότι θα δηλώσει ότι θα είναι νόμιμο να, περάν, να περνά τα σύνορα αυτά τα φορτικά πριν ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου επίσης ε, θα γνωμοδοτήσει για να δούμε αν έχει την ίδια άποψη με την Κομισιόν. Ε, Εν τω μεταξύ, μίλησα με τον κύριο Επίτροπο, μου είπε σήμερα το πρωί πως δεν θα γίνει καμία ανακοίνωση για τα φορτίγα αυτά. Και αυτό οπωσδήποτε δεν θα γίνει πριν έρθει ο κύριος Κάλλας να μιλήσει στην Επιτροπή μας για τις προθέσεις του. Οπότε όσον αφορά την διαδικασία που ανησυχούσε πολλούς βουλευτές, ο κύριος Κάλλας θα έρθει στο Κοινοβούλιο, θα εξηγήσει την απόφασή του και οπωσδήποτε τότε Έγινε μια συζήτηση έντονη και εις βάθος μεταξύ των μελών της Επιτροπής και του κυρίου Κάλλας σε σχέση με την απόφαση αυτή. Αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε πως στην αρχή ανησυχούσα και εγώ, όπως και οι συντονιστές, πως αυτό θα γινόταν χωρίς ε, καμία συνεννόηση με το Κοινοβούλιο. Αυτό το είπαμε και οπωσδήποτε το δέχτηκε ο Επίτροπος και θα έρθει στο Κοινοβούλιο να δώσει εξηγήσει για το τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με τα τεράστια φορτηγά πριν κάνει οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Ζητήθηκε από τον πρόεδρο να ζητήσει από την Κομισιόν περισσότερες πληροφορίες για το πιο ποιοι εσωτερικοί λιμένες συμπεριλαμβάνονται στα προτινόμενα δίκτυα το βασικό και το εκτεταμένο. Γιατί υπάρχει κάποια σύγχυση σε σχέση με το ποιοι ε, λιμένες εσωτερικής ναυσικλωίας περιέχονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και στο βασικό και εκτεταμένο δίκτυο. Θα ζητήσουμε λοιπόν διευκρινήσεις. Επίσης, έγινε μια συζήτηση για την ποιότητα του αέρα στα αεροσκάφη που το έθεσε ο κύριος Κράμερ ε, εξ των Πρασίνων και αποφασίσαμε να ασχοληθεί ο κύριος Κράμερ με το θέμα να ρωτήσει την Κομισιόν και να ενημερώσει τους συντονιστές όταν ε, το απαντήσουν από την Κομισιόν και από άλλες πηγές για να μπορούν μετά οι συντονιστές να ξαναδούν το θέμα. Νομίζω αυτά είναι όλα. Ο κύριος Κοχ επίσης για, ε, ε, για το οίκο με το οποίο θα ασχοληθεί. Λοιπόν, Φαντάλεν, Λίχτενμπέργκερ, Λάιχτφριντ, Κοχ, Κάντσιαν, θα λάβουν όλο το λόγο για αυτά που σας είπα για τους ε, συντονιστές. Αν μπορείτε λοιπόν να είστε σύντομοι, θα σας ήμουν ευγνώμων. κύριος Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Εγώ είμαι ικανοποιημένος ε, με την θέση του Επιτρόπου Σάλας για τα φορτηγά αυτά. Ε, δεν μπορούσα, δεν θα περιμένω τίποτα άλλο. Πάντα έρχεται ο κύριος Κάλλας εδώ πέρα και μας ακούει και συνεργάζεται μαζί μας. Υπάρχει λοιπόν σαφήνεια, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω και εσάς και τους συναδέλφους να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πρόκειται για φορτηγά, με μεγαλύτερα και βαρύτερα φορτηγά. Οι λοιποί όροι που χρησιμοποιούνται δεν είναι σωστοί και οι εμπειρίες που έχουμε στην Ολλανδία είναι μόνο θετικές ε, και όσον αφορά την οδική ασφάλεια και όσον αφορά και την κυκλοφορία. Οπότε σας παρακαλώ να χρησιμοποιείτε τους όρους μεγαλύτερα και βαρύτερα φορτηγά. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ μην μπείτε σε συζήτηση για τα φορτηγά τώρα. Μείνετε σε αυτά που σας είπε ο Πρόεδρος. Κύριε Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ. να κάνω ένα σχόλιο για τον ε, κύριο Μπρίνκχορστ, τον συντονιστή των διευρωπαϊκών δικτύων και τον Λεόν Τουρίν, μαζί με τους ε, για την υπόθεση της σύνδεσης με το, το Φαίνεται πως υπάρχει μία ε, έλλειψη πληροφόρησης για το θέμα Επίσης για τους εσωτερικούς ε, λιμένες και το μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη. Εάν μιλάμε και για τους θαλάσσιους ε, λιμένες, αν είναι αντί να μην κάνουμε απλά μια απαρίθμηση, αλλά να έχουμε κάτι το, το χρήσιμο, γιατί ξέρετε στον Νότο δεν έχουν τεθεί προτεραιότητες γιατί νομίζω πως ε, θα μπορούσαμε να δώσουμε και προτεραιότητες ε, και στα ε, λιμάνια. Εάν είναι πράγματι να δώσουμε ένα μεγαλύτερο βάρος και να ενσωματωθούν καλύτερα αυτά στην εργασία μας. Γιατί ξέρετε πως όταν είχαμε κάνει ακριβώς τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου είχαμε πει πως θα δοθεί προτεραιότητα ακριβώς στα λιμάνια, όχι μόνο στους εσωτερικούς λιμένες και στους ε, υπόλοιπους. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο μία παρήθμιση. Σας ευχαριστώ. Το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω είναι να σας πω εγώ το τι ε, συζητήσαμε οι συντονιστές. Μιλήσαμε ειδικά για τους εσωτερικούς λιμένες. Αν θέλετε να το προχωρήσετε βεβαίως μπορείτε. Δεν λέω αν έχετε δίκιο ή άδικο, αλλά το συγκεκριμένο θέμα που συζητήσαμε και έτοιμα αφορούσε την εσωτερική ναυσιπλογία. Λοιπόν, ο κύριος Λάχιφεριτ. Ευχαριστώ. Για τα φορτηγά, τα, τα τεράστια. Τέσσερα, τώρα δεν θέλω να αντιπαρατεθώ με τον Πίτερ επί της ουσίας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πως υπάρχει ένα ισχύον δίκαιο πριν από λίγα χρόνια από το Συμβούλιο αποφασίσαμε το τι θα γίνει. Ότι τα κράτη-μέλη με τη σύμφωνη γνώμη της ε, Κομισιόν μπορούν ή ε, να επιτρέψουν ή όχι στην επικράτειά τους τα φορτηγά αυτά. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι ξεκάθαρη παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ωραίο είναι να έρθει εδώ πέρα ο κύριος Επίτροπος να μας πει γιατί παραβιάζει το δίκαιο, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν είναι να υπάρξει κάποια αλλαγή θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία. Πρόταση δηλαδή της Κομισιόν για να αλλάξει αυτή η οδηγία και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Αλλά δεν γίνεται έτσι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Επίτροπος, ο Επίτροπος, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποτίθεται πως είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων να το παραβιάζει. Το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όχι, δεν γίνεται. Ανεξαρτήτως του αν είναι καλό ή κακό επί της ουσίας. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά όσο είναι το δίκαιο αυτό που είναι, δεν μπορεί να το παραβιάζει η Κομισιόν. Όπως μου λέει και η Επίτροπος ε, κυρία Χέντεγκαρτ συχνά, ο νόμος είναι ο νόμος. Τώρα, μίλησα στον Επιτρόπο, του ξεκαθάρισα τι ε, απόψει μα. Ανεξαρτήτως του αν είναι καλά ή κακά αυτά τα φορτηγά, τα τεράστια, όλοι έχουμε τι απόψει μα. Εγώ συμφωνώ περισσότερο μαζί σα παρά με κάποιου άλλου βουλευτέ. Πράγματι, πράγματι ο κύριο Φαντάλεν έχει διαφορετική άποψη. Και δεν, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ ανισχώ με την ε, κυριαρχία του Κοινοβουλίου και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Γι' αυτό για μένα σωστό ήταν να έρθω σε επαφή με τον Επίτροπο να του πω πως δεν με ικανοποιεί αυτή η διαδικασία το ότι πρώτα απ' όλα υπήρξε μια διαρροή μετά θα ε, ε, υπήρχε μια ανακοίνωση στην ε, Διεθνή Ένωση Μεταφορών προφανώς έχει λάβει το μήνυμα τώρα πως θα πρέπει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο πριν ε, ανακοινώσει πως υπάρχει κάποια αλλαγή στην ε, πολιτική. Γι' αυτό, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπατε κύριε Λάιχτριντ, πρέπει να έχουμε κι εμείς δική μας νομική γνωμοδότηση. Έχουμε τη γνωμοδότηση της ε, Κομισιόν που λέει πως είναι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, υπό την υφιστάμενη νομοθεσία, τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν την διασυνοριακή κίνηση των φορτηγών αυτών ε, στην επικράτειά τους. Οπότε είναι θέμα επικουρικότητας, αλλά χρησιμοποιούν ε, την υφιστάμενη νομοθεσία και μια νέα ερμηνεία. Όπως ξέρετε, δεν είμαι δικηγόρος, ε, δεν είμαι νομικός. Οπότε, οι συντονιστές λένε πως χρειαζόμαστε δική μας μια άλλη γνωμοδότηση. Νομίζω σωστό είναι αυτό. Γιατί ο κύριος Κάλλας θα έρθει και θα μας πει ποια είναι η απόφαση του και δεν θα ανακοινώσει τίποτα άλλο και ξέρουμε ποια είναι η απόφαση. Οπότε έχουμε χρόνο ε, έτσι ώστε και η δική μας νομική υπηρεσία να το δει. Ε, συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, πράγματι ο ρόλος μου, εμένα ως πρόεδρος, ανεξαρτήτως της άποψής μου επί της ουσίας, είναι ακριβώς η κυριαρχία του Κοινοβουλίου και το ότι δεν ε, ζητήθηκε η γνώμη μας για μια ριζική αλλαγή στην πολιτική. Και αυτό οπωσδήποτε το, το τόνισα. Ναι, ναι, σύντομα. Ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, θα είναι τακτική συνεδρίαση, θα είναι μια πληροφόρηση των συντονιστών. Εύα, είναι 9.30 ώρα, ε, 9 ε, παρά με πήραν τηλέφωνο. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Υποθέτω, απαντά ο πρόεδρο σε μια ερώτηση που δεν ακούστηκε, γιατί πρέπει να το κανονίσουμε και χρειαζόμαστε χρόνο και εμεί και η Κομισιόν για να το σκεφτούμε. Ο κύριο Κάντσιαν. Ευχαριστώ. Εντάξει, σε σχέση με το ΣΤΟΑ, εμείς είχαμε δύο αιτήματα, δύο εκθέσεων, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αυτό που με απασχολεί είναι η προθεσμία της 8ης Μαΐου. Ακόμα βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο. Τι θα γίνει με την ακρόαση των τεν t και των, του μέσου. Το θέμα αυτό διαρκεί πάρα πολύ και του μέσου Connecting Europe. Εάν για το Connected Europe είναι εντάξει, γιατί μιλάμε για το 14-20, για το TEN-T νομίζω ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε. Γιατί ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε θέματα χρηματοδότησης. Εάν ισχύσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός από εμάς. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να την ε, απομακρύνουμε από το CEF, από το μέσο Connecting Europe. Δηλαδή να αποχωριστούν το ένα από το άλλο. Γιατί άλλο είναι το μέχρι 13 και άλλο 14 με 20. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς έχει η πρόταση που μας έκανε η Επιτροπή. Αντώνιο. Ναι, το έχω επιταχύνει το μέσον Connecting Europe είναι ε, πρώτο γιατί πρέπει να λήξει τον Απρίλιο και τώρα είμαστε στις αρχές Μαρτίου. Δεν μπορούσαμε να επιταχύνουμε γιατί έχουμε το Πάσχα το οποίο υπησέρχεται. Μιλάμε και για το καθολικό και για το ορθόδοξο Πάσχα, τα οποία δεν συμπίπτουν. Δεν ήξερα ποτέ ότι θα γίνω η Δήμον για το Πάσχα και τη διαφοροποίησή του, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι αίθουσε έχουμε, ποιου εμπειρογνώμονε μπορούμε να καλέσουμε. Η 8η Μαΐου θα φτάσει ε, νωρίτερα από όσο φανταζόμαστε και από ό,τι βλέπουμε από τους εισηγητές δεν θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, άρα έχουμε χρόνο. Το εκτιμώ. Είναι σημαντικό. Πολλά συμβαίνουν στα κράτη-μέλη, με φορείς, οργανώσεις και ούτω καθεξής, αλλά νομίζω ότι η 8η Μαΐου είναι η πρώτη εφικτή ημερομηνία που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το δούμε μαζί με το ΣΕΦ. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται με το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Άρα σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Θα κινηθούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Προσπαθώ να το δούμε το συντομότερο. Κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συμμερίζομαι απολύτως την, ε, τον προβληματισμό του συναδέλφου για γρήγορες κινήσεις στο θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Όμως, και αυτή ήταν και η προσπάθεια και η δική μου και ε, του κυρίου Ερτούγκ, να έχουμε το συντομότερο δυνατόν μια, ε, ένα public hearing για αυτό το θέμα. Για διαδικαστικούς και άλλους λόγους στους οποίους αναφερθήκατε, δεν έγινε εφικτό. Και εγώ θα ήθελα και η προσπάθειά μας ήταν να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε εφικτό και έτσι πάμε για, τις, ε, για την 8η Μαΐου παρά το γεγονός ότι θα προτιμούσαμε να ήταν πολύ νωρίτερα. Ευχαριστώ. Indeed, I, dealing with... Ως προς τις ε, διαδικασίες του Κοινοβουλίου, εσείς που έχετε βρεθεί σε αυτή τη θέση, ξέρετε ότι αυτός ο γκόλιθος που λέγεται Κοινοβούλιο είναι ένα δύσκολο θέμα πώς θα το διαχειριστεί κανείς. Κόχ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω κάτι θετικό για τα φορτηγά. Τέλος πάντων, δεν τα αφήνω. Απλά θα ήθελα να πω κάτι άλλο για τα βιοκαύσιμα τα οποία θέτε να, να μετονομάσετε σε αγροκαύσιμα. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται κατά βάση για οργανικά απόβλητα και άρα έχουν ένα θετικό οικολογικό αντίκτυπο. Μάλιστα, θα πρέπει να, τώρα θα πρέπει να δούμε τον ορισμό βιοκαυσίμων και αγροκαυσίμων. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Κυρία Φώστερ. Δεν θα μιλήσω για το θέμα των καυσίμων. Ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος ε, Κράμερ, για την ποιότητα του αέρα μέσα στα αεροπλάνα, ε, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό λόμπι το οποίο προσπαθεί να επικρατήσει. Εγώ δεν είμαι επιστήμον, άρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Ξέρω ότι σε ορισμένα αεροσκάφη στο παρελθόν κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτά τα συστήματα εξαερισμού. Αλλά πέρα από αυτό, με ποιον θα ε, έρθετε σε επαφή. Από ποιους θα λάβετε πληροφορίες σε σχέση με αυτό το θέμα. Κανέναν, λέει ο πρόεδρος. Οι συντονιστές αποφάσισαν ο κύριος Κράμερ να έρθει με αποδεικτικά στοιχεία για να δούμε τι θα κάνουμε. Άρα αυτή τη στιγμή η άποψη των συντονιστών ήταν να μην κάνουμε κάτι το συγκεκριμένο. Θα περιμένουμε από τον κύριο Κράμερ να μας φέρει στοιχεία από τα συνδικάτα, από άλλους φορείς και μετά θα επανέλθουμε στους ε, συντονιστές για να ορίσουμε κάτι το συγκεκριμένο. Τότε δεν κατάλαβα καλά, γιατί όταν έγινε αναπομπή Είπατε ότι θα, θα το ερευνήσουμε. Ο κύριος Κράμερ θα το κάνει αυτό, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα ως προς τους συντονιστές και τις ανακοινώσεις του Προέδρου, την εισήγηση του Προέδρου, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Τώρα προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η δική μου έκθεση για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και η παρουσίαση της έκθεσής μου. Η πρόταση της Επιτροπής είναι να μεταφέρουμε τις αλλαγές που ήδη συμφωνήθηκαν από τα κράτη-μέλη στην σύμβαση STCW του IMO έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με το STCW με την σύμβαση αυτή για την εκπαίδευση των ναυτικών. Γι' αυτό η εμβέλεια των αλλαγών είναι πολύ μικρή, πολύ περιορισμένη. Οι προηγούμενες ε, τροποποιήσεις έχουν ήδη μεταταχθεί στην κοινοτική ένωμη τάξη με παρόμοιες οδηγίες. Εγώ Ζήτησα να λάβουμε υπόψη την τροποποίηση Μανίλα έτσι ώστε για λόγους αφήνειας να επικαιροποιήσουμε το κείμενο ανάλογα με τις πρόσφατες ε, εξελίξεις. Εκεί που έγιναν αλλαγές ε, αφορούν το εξής οι αλλαγές. Ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις περιόδους ανάπαυσης και για τις ασκήσεις όσον αφορά τις νέες απαιτήσει της ε, προτινόμενης οδηγίας, πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένε λεπτομέρειε όσον αφορά τα πιστοποιητικά κατάρτιση των ναυτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αιτήσια βάση, προκειμένου να υπάρχει μια πιο σφαιρική εικόνα του επάγγελμα του ναυτικού στην Ευρώπη. Ως προς αυτό θα ήθελα να επιφέρω τις εξή ε, αλλαγέ θα ήθελα να προστατεύσω περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα των ναυτικών, ζητώντας να είναι ανώνυμα τα δεδομένα αυτά που θα δίδονται για τους ναυτικούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει όρος anonymization, το οποίο χρησιμοποιήσει στο αγγλικό κείμενο. Ουσιαστικά θέλουμε να είναι ανώνυμοι ναυτικοί, των οποίων τα δεδομένα θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θα πρέπει τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, να εξασφαλίσουμε επίσης ότι τα στατιστικά στοιχεία που θα εφίστανται επεξεργασία θα είναι διαθέσιμα στο κοινό και επομένως υποστηρίζω στεναρά τη συλλογή δεδομένων για το επάγγελμα του ναυτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει σαφής ανάγκη για πληρέστερη εικόνα της κατάστασης απασχόλησης στον λόγο τομέα. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της αναθωρημένης επιτροπολογίας, Έχω χρησιμοποιήσει μια νέα διατύπωση προκειμένου να αντικατοπτρίσετε καλύτερα το διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 όσον αφορά τις κατεξοδότηση πράξης. Επίσης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διακρίσεις ανάμεσα στα πιστοποιητικά α, ικανότητας και επάρκειας, έχω επιφέρει επίσης κάποιες τροποποιήσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τροποποιήσεις της Μανίλα άρχισαν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Δεν θα πρέπει λοιπόν να καθυστερήσει περισσότερη η ευθυγράμμιση της κοινοτική νομοθεσίας με τις απαιτήσει των τροποποιήσεων της Μανίλα. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σύγκρουση ανάμεσα στις υποχρεώσεις τις κοινοτικέ και τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη ως μέρη της συμφωνίας της ε, τη συμφωνία STCW. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί πολύ γρήγορα μία συμφωνία. Έχω κάνει λοιπόν κάποιες τροποποίησεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω ότι οι τροποποίησεις αυτές θα γίνουν αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, εργάστηκα πολύ στενά με τον κύριο Όλε Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι ο εισηγητής για την γνωμοδότηση που θα κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης όσον αφορά κάποιες αλλαγές που γίνονται στα άρθρα τα οποία θέτουν τις εξαιρέσεις για τις ελάχιστες ε, ε, ώρες ανάπαυσης. Και εδώ πέρα οι τροποποίησεις της Μανίλα ουσιαστικά είναι ε, πιο ήπιε από αυτέ που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία. Προσπαθώ λοιπόν να συνεργαστώ με τον συνάδελφό μου από την Επιτροπή Απασχόληση, προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία και με την Δανέζικη Προεδρία για το ζήτημα αυτό και προκειμένου να καταφέρουμε ομαλά να περάσουμε τις τροποποίησεις της Μανίλας στην κοινοτική νομοθεσία το συντομότερο δυνατό. Αυτά είχα να σας πω, κύριος Κουμουτσάκος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης έχει στρατηγική σημασία για την διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια ναυτιλία. Επομένως, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης είναι ένας βασικός παράγοντας που πρέπει <clears throat> να στηρίξουμε. Παρά το γεγονός ότι είμαστε σε εποχή οικονομικής δυσκολίας, η ναυτική εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται κόστος αλλά επένδυση. Άλλωστε, βελτιώνει την ελκυστικότητα των ναυτικών επαγγελμάτων και βέβαια την ασφάλεια ε, και την προστασία της ναυσιπλοείας. Ε, γι' αυτό καλωσορίζω και εγώ την ε, πρόταση της Επιτροπής για την, για την τροποποίηση της προηγούμενης οδηγίας ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τα όσα αποφασίστηκαν στην Συμφωνία της Μανίλας το 2010. Οι τροπολογίες σας, κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητού κινούνται σωστή κατεύθυνση. Ε, ειδικά θέλω να υποστηρίξω την πρότασή σας για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων των ναυτικών και ε, βεβαίως να τονίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία που θα δίδονται από τα κράτη-μέλη προς την Επιτροπή θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να θίξω, τα οποία νομίζω ότι αξίζουν προσοχή. Το ένα αφορά την έναρξη ισχύω της οδηγίας την οποία ξεκινήσαμε να συζητάμε. Σε σχέση με τον χρόνο ισχύω, με την έναρξη ισχύω τη Συμφωνία τη Μανίλα. Η Συμφωνία τη Μανίλα προβλέπει έναρξη ισχύω την 1η Πρώτου του 2012, δηλαδή ουσιαστικά έχει αρχίσει η ισχύ τη, ενώ η δική μα ε, νομοθετική διαδικασία θα φτάσει να <clears throat> ισχύει η, η, η οδηγία τουλάχιστον 6-7 μήνες μετά. Στο μεσοδιάστημα δημιουργείται ένα πρόβλημα. Τα καράβια, τα πλοία με σημαίε ευρωπαϊκές των κρατών μελών θα πρέπει είτε να συμφωνήσουν με τη Διεθνή Σύμβαση εφόσον την κυρώσουν και έτσι να μην συμφωνούν με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο είτε να μην την ε, κυρώσουν περιμένοντας τη δική μας οδηγία να ε, τεθεί σε ισχύ και έτσι να είναι έκθετα σε τρίτα κράτη με τα οποία συνεχίζουν να έχουν εμπορικές συναλλαγές και τα οποία τρίτα κράτη έχουν ήδη κυρώσει και εφαρμόσει ε, τη Μανίλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο, ε, κύριε Πρόεδρε, αλλά σίγουρα πρέπει να κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν για να προχωρήσουμε και να κλείσουμε αυτήν την ε, οδηγία την οποία συζητάμε σήμερα. Ενδεχομένως να υπάρχει κι άλλος τρόπος να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, αλλά δεν το γνωρίζω. Εδώ <clears throat> αυτό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η ανάγκη ταχύτητας. Και ένα, δεύτερο και τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε στο συγκεκριμένο κείμενο καινούργια στοιχεία, διότι ουσιαστικά πρόκειται για μια προσαρμογή και μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο της Συμφωνίας Μανίλας. Όμως, υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και ιδιαίτερη. Είναι η εκπαίδευση των ναυτικών στην αντιμετώπιση περιστάσεων και περιπτώσεων πειρατείας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι πράγματι το φαινόμενο είναι μια πραγματική μάστιγα και θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να μπει κάτι σε αυτό το κείμενο και εν πάση περιπτώσει εγώ θα καταθέσω μια τροπολογία είτε ως άρθρο είτε ως recital για την ανάγκη να υπάρξει πρόβλεψη εκπαίδευση των ναυτικών, κατάλληλη εκπαίδευση και για την αντιμετώπιση περιστάσεων πειρατεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τα άλλα θα, καταθέ, θα κατατεθούν ως τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενο, γιατί παρά το γεγονός ότι δεν έχει πολύ μεγάλη πείρα επί του θέματος, μπόρεσε να συνεισφέρει σε αυτό το θέμα επί της ουσίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε και να δούμε να λάβουμε υπόψη και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια ελιγμών για να μπορέσουμε να αναδιατυπώσουμε τις προγενέστερες οδηγίες σε σχέση με την πιστοποίηση των ναυτικών. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής στην ουσία προσαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με τις αλλαγές που έχει επιφέρει η ΙΜΟ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κείμενο του κυρίου Σίμψον στην ουσία βελτιώνει το κείμενο, είναι πιο επεξηγηματικό και πιο σαφές. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ενίσχυσης προσωπικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς, εκεί όπου υπάρχει υποχρέωση ανωνυμίας. Έτσι, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να δημοσιεύουν τα στοιχεία, αλλά παράλληλα θα υπάρχει η εγγύηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα. Υπ' αυτή την έννοια, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία για όλα τα επαγγέλματα του κλάδου. Και αυτό θα έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στο ίδιο το επάγγελμα. Και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την ανεργία η οποία διέπει τον τομέα αυτή τη στιγμή. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μείνει πίσω. Το είπε και ο πρόεδρος Σίμψον και ο κύριος Κουμουτσάκος. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία, διότι η σύμβαση της Μανίλα ε, στην ουσία ε, κυρώθηκε το 10, ενώ άρχισε να ισχύει την 1η του 12. Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε επίσης για την διεξοδική παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Υποστηρίζουμε εν γέννη τα όσα προσπαθείτε να κάνετε. Είναι σαφές, είναι προφανές, το ότι χρειαζόμαστε την κατάλληλη εκπαίδευση για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα αυτό, για τους ναυτικούς, και πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτό. Νομίζω ότι αναφερθήκατε στα βασικότερα σημεία. Μία βασική ανησυχία που έχουμε εμείς είναι ότι όταν εξετάζουμε την μεταβίβαση δεδομένων από μία βάση δεδομένων σε ένα κράτος μέλος προς μία άλλη βάση δεδομένων, της ΕΜΣΑ για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει απόλυτα μία συμμόρφωση στα συστήματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα κράτη-μέλη όταν θα χρειαστεί να μεταβιβάσουν, να διαβιβάσουν αυτές τις πληροφορίες. Να δούμε δηλαδή και ποιο θα είναι το χρονικό πλαίσιο της διαβίβασης των δεδομένων. Θα πρέπει το χρονικό αυτό πλαίσιο να είναι ρεαλιστικό, προκειμένου τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση. Κάτι άλλο σημαντικό που είπατε έχει να κάνει με την ε, ανωνυμία των ε, δεδομένων. Δεν ξέρω ακριβώ και ποιο είναι αυτό ο όρο που χρησιμοποιείται στα αγγλικά. Έχετε πάντω δίκιο. Και νομίζω ότι η σχετική τροπολογία όντω ε, αντανακλά την ανάγκη αυτή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε προσωπικά δεδομένα, προσωπικέ λεπτομέρειε για του ανθρώπου αυτού να είναι διαθέσιμα παντού. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ενισχύσατε το σημείο αυτό και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το λάβει αυτό υπόψη. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ο εμπιστευτικό χαρακτήρα είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη του σα. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αποτελεί το κέντρο διαμόρφωσης των διεθνών κανόνων για την αυθυλία, συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής εκπαίδευσης, γενικότερα των κανόνων για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος. Συμφωνώ με την εκτίμηση την άποψη του εισηγητή ότι η πρόταση της Επιτροπής συνίσταται κυρίως σε άσκηση μεταφοράς των αλλαγών που έχουν ήδη συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη στη Σύμβαση της STCW του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με σκοπό να ευθυγραμμιστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με την τροποποιημένη σύμβαση και τις αλλαγές που περιέχονται. Επιτρέψτε μου όμως εν συντομία να κάνω ορισμένες εκτιμήσεις τάχει. Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία σε ό,τι αφορά το τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες που υπάρχουν τόσο στο επίπεδο μεταξύ των 100 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μεγαλύτερη έκταση των 100 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Και αυτό συνίσταται το ότι ενώ τα 34 τελευταία χρόνια η εφαρμοσμένη τεχνολογία στα πλοία έχει αυξηθεί με σύγχρονα πλοία, με σύγχρονο εξοπλισμό, αυτό δεν έχει περάσει στους ναυτεργάτες που χειρίζονται και δουλεύουν στα πλοία. Α, επιπρόσθετοι παράγοντες που πραγματικά αποτελούν μεγάλο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την διεθνή ναυσιπλοεία, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, είναι ότι έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί ο χρόνος φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ταχύτητα των πλοίων, έχουν μειωθεί οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων, και προφανώς είναι θετική η πρόταση που γίνεται από τον εισηγητή σε ότι να εξασφαλιστούν έστω τα ελάχιστα όρια ανάπαυσης σε ό,τι αφορά για τους ναυτεργάτες των πλοίων και κατά τη διαδικασία των ασκήσεων. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να επισημάνω ότι όχι μόνο καταστατηγούνται αλλά και αυτά τα μέτρα που ποτείνονται δεν πρόκειται να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Έτσι ε, επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση, τροπολογία, στα πλαίσια της δυνατότητας που υπάρχει και δίνεται σε ό,τι αφορά τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, αφού, όπως πρέπει να ίσως να ξέρετε, οι περισσότεροι, το προσωπικό ενδιέτησης των πλοίων, δηλαδή όλο το προσωπικό που ιδιαίτερα στα κουραζερόπλια μπορεί να αποτελεί και εκατοντάδες κατά πλοίο, κατά μονάδα πλοίου, δεν θεωρείται μέλος της οργανικής σύνδεσης των πλοίων. Και για, αυτά το, και για αυτό το προσωπικό δεν περιλαμβάνεται στους κανόνες και στους όρους ανάπαυσης. Να τελειώσω με το εξής. Έχουμε την παλαιότερη πείρα της, κωδικοποίηση της κωδικοποίησης της ναυτεργατικής νομοθεσίας ε, του 2006 από τη Διεθνή Οργάνωση ε, Εργασίας. Ε, με την πρόφαση να συζητηθεί μέσα στα εσωτερικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα τρία επίπεδα, Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάθηκε πολύς χρόνος, απονευρώθηκαν πολλά στοιχεία θετικά από αυτή την νομοθεσία, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι αυτό που κατά την άποψή μας προτείνουμε είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έστω να υλοποιηθεί άμεσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα η συγκεκριμένη ε, πρόταση της SCCW για την ναυτική εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Mrs. Vlasto. Κύριε Βλαστό, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφό μου τον Γιώργο, για την καταπολέμηση της πειρατείας δηλαδή. Όπως είπες και εσύ, θα ήθελα και εγώ να υπάρχει κατάλληλη ειδική εκπαίδευση για τους ναυτικούς, για το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στον κώδικα καλής συμπεριφοράς που υπάρχει σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Δεν υπάρχει λόγος να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό από την αρχή. Νομίζω ότι μας κάνει πάρα πολύ αυτό το οποίο υπάρχει στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρο ότι κατάλαβα πολύ καλά. Όσον αφορά τις ε, ασκήσεις εκένωσης ή τις ασκήσεις για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμφωνείτε να μην ενσωματωθούν στην περίοδο ανάπαυσης, να μην... γιατί καταλαβαίνετε ότι στην περίοδο αυτή, στην, στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να πρέπει κανείς να πρέπει να κάνει ασκήσεις ενώ τη στιγμή εκείνη προβλεπόταν μια περίοδος ανάπαυσης. Η περίοδος ανάπαυσης είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε πρόκειται για τις οδικές μεταφορές, είτε πρόκειται για τις αεροπορικές μεταφορές και νομίζω ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και τις θαλάσσιες μεταφορές. Καραμίτσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη της Επιτροπής σας. Νομίζω ότι όλοι λέτε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία, ότι θα πρέπει να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο, προκειμένου να αρχίσει να ισχύει η νομοθετική αυτή πράξη. Γιατί όντω μιλάμε κυρίω για μια μεταφορά διεθνού δικαίου. Βλέπουμε ποιε είναι οι απόψει σας ότι ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα της ε, προστασίας των δεδομένων. Σε ζητώ συγγνώμη για τον αγγλικό αυτό όρο που χρησιμοποιούμε. Εμείς πολλές φορές ε, δημιουργούμε εδώ πέρα όρους που μπορεί αργότερα να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται για την περίοδο ανάπαυσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα πούνε και οι συναδελφοί από την Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά με τη δική σας συνεργασία και με την Προεδρία θα προσπαθήσουμε και γι' αυτό να βρούμε μια καλή και γρήγορη λύση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί, να τηρηθεί προφανώς. Ένα ζήτημα το οποίο ανέφερε ο κύριος Κουμουτσάκος νομίζω και η κυρία Βλαστό είναι το ζήτημα της πειρατείας. Όντω υπάρχουν στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού κάποιες σχετικές συστάσεις. Δεν καλύπτουν όμως το ζήτημα της σχετικής εκπαίδευσης. Μιλάμε κυρίως για βέλτιστες πρακτικές, πώς θα πρέπει να αντιδράσει κανείς σε περίπτωση επίθεσης, πώς θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο το πλοίο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασιζόμενη στις συστάσεις αυτές έχει κάνει τις δικές της συστάσεις. Τώρα όμως η σχετική εκπαίδευση για την καταπολέμηση της πειρατείας, ναι, αυτό θα μπορούσαμε στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να το λύσουμε και να βρούμε και μια σχετική διατύπωση σε κάποιο εκτιμώντας στην αιτιολογική σκέψη του κειμένου. Θα μπορούσατε και εσείς να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια αναφορά στο ζήτημα αυτό. Πάντως δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το νομοθετικό αυτό, το νομικό αυτό κείμενο προσθέτοντας κάτι σχετικό. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, δεν υπάρχει το ζήτημα αυτό ακόμα στην ατζέντα εργασίας του Συμβουλίου, αλλά μπορούμε και αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Ένα ακόμα ζήτημα, λίγο πιο θεσμικό, έχει να κάνει με την εφαρμογή των κατεξοδότηση πράξεων. Υπάρχει το νομικό τμήμα και το τεχνικό, αν θέλετε, τμήμα του όλου ζητήματος. Στο παρελθόν, στα πλαίσια της ε, σύμβασης STCW, προσπαθούσαμε να περάσουμε στην κοινοτική νομοθεσία οποιασδήποτε τροποποίησεις γινόντουσαν και τροποποίησεις που είχαν συζητηθεί ακόμα και στην ΕΜΣΑ. Δεν νομίζω ότι ε, θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα αν καθυστερήσουμε λίγο τη διαδικασία λήψης απόφασης, αλλά θέλουμε και εμείς να διατηρήσουμε την ε, διοργανική συμφωνία και να βρούμε μία λύση. Είμαστε πάντως σε θέση να σας βοηθήσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις βελτιώσεις που έχετε προτείνει για το νομικό τμήμα του κειμένου. Σχετικές τροποποιήσεις, βελτίωση έχουν γίνει και από το Συμβούλιο και ελπίζω ότι πριν το καλοκαίρι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για το κείμενο αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να λάβω το λόγο σε σχέση με αυτά που είπαν τα μέλη πολύ χρήσιμα θέματα για την εκπαίδευση των ναυτικών, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει περισσότερο. Δεν διαφωνώ με κάτι, με όσα προελέχθησαν από τους Τούσα και Βλαστό. Το ζήτημα είναι ότι έχω να κάνω με ένα κείμενο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Και αν και θα ήθελα να μπορέσω να αλλάξω τους κανόνες του IMO, δεν μπορώ και να θέλω δηλαδή και σας εκπλήσει αυτό. Το μόνο λοιπόν που μπορώ να κάνω είναι να μεταφερθεί πρωτίστως στο κείμενο και μετά μπορώ να το τροποποιήσω εκεί όπου πληττόμεθα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτροπολογία, προστασία δεδομένων και ούτω καθεξής. Σε αυτούς τους τομείς και μόνο. Σε σχέση με το θέμα που είπε ο κύριος ε, Κουμουτσάκος για την εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση πειρατείας, βεβαίως μπορεί να την αναλάβει οποιοδήποτε. Αλλά δεν υπάρχει στο κείμενο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού κατά πόσο πρέπει να κάνει περισσότερα ο IMO. Ε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και ο κύριος Φλέκενστάιν έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια της ΕΜΣΑ και γι' αυτό νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την ε, πειρατεία. Γιατί εδώ μιλάμε μόνο για μεταφορά των οδηγιών. Κάνω λοιπόν αυτή την έκκληση. Ο κύριος ε, Τούσας είπε ότι θα υποβάλει τροπολογίες για την εκπαίδευση. Δεν ξέρω κύριε Τούσα κατά πόσο θα επιτραπούν γιατί από νομικής πλευράς εμείς μεταφέρουμε ένα κείμενο του Διεθνούς ε, ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού. Καταλαβαίνω απόλυτα τι προσπαθείτε να κάνετε και δεν σημαίνει ότι αντίκειμε αλλά χρειαζόμαστε να πιέσουμε τον IMO για καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερα πρότυπα και προδιαγραφές. Ως προς αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα, ως προς τις ασκήσεις, κυρία Βλαστό. Αν χρειαστόμαστε ασκήσεις, να το βλέπουμε και στο Κώστα Κονκόρδια, που δεν έγιναν ασκήσεις εκένωσης. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης να υπάρχουν και αυτές οι ασκήσεις. Αυτό είναι το θέμα μας μέσα στα πλαίσια της μετάταξης των διατάξεων του IMO. Αυτά είναι τα θέματα που θέλω να θίξω σε σχέση με αυτά που είπατε εσείς. Κάνω μια έκκληση. Σας λέω ότι αυτό δεν είναι έκθεση που ορίζει προδιαγραφές εκπαίδευσης για τους ναυτικούς. Δεν είναι. Δεν είναι. Μιλάμε για μεταφορά της νομοθεσίας του IMO στην εσωτερική ένωμη τάξη μας. Είπατε ότι είμαστε, έχουμε μείνει πίσω. Έχετε πολύ, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό γίνεται εξαιτία του Ευρωπαϊκού Συνομιλίου. Διότι η Επιτροπή Απασχόλησης είπε να ισχύσει το άρθρο 50. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κοινή έκθεση. Εμείς το αμφισβητήσαμε αυτό και αυτό οδήγησε σε χρονοτριβή και σε καθυστέρηση. Η ε, Δανική Προεδρία ήθελε ήδη να το προωθήσει, αλλά αυτός αυτό το γελίο άρθρο προκάλεσε την καθυστέρηση. Δηλαδή, δυστυχώς, εμείς είμαστε υπέτη της καθυστέρησης. Δεν φταίει ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Επιτροπή, ούτε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Εμείς φταίμε αποκλειστικά. Ωραία. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 22 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω όμως, από τεχνικής πλευράς, ξέρετε, ξέρετε. Μιλάμε για μεταφορά μόνο. Τον Απρίλιο θα ψηφίσουμε και είτε τον Μάιο είτε τον Ιούνιο θα ψηφίσει ολομέλεια. Για το θέμα αυτό, για την εκπαίδευση, για την πειρατεία, το δέχεστε ως ένα εκτιμώντας κάπου, να μην αλλάξει το διατακτικό, ως εκτιμώντας ίσως. Ναι, ε, Σκέφτομαι μεγαλοφόνο Το πρόβλημα είναι πως μπορεί να έρθει ο κύριος Τούσας μετά και να μας πει δεχτείτε και όλα αυτά σαν εκτιμώντας. Και ανησυχώ με, μην ανοίξουμε έτσι το κουτί της Πανδώρας. Η πρότασή μου κύριε Κουμουτσάκο είναι ε, θεμητό αυτό που λέτε αλλά ίσως καλύτερα να πάει στην έκθεση του κύριου Φλακενστάιν για την έμψα αντί για αυτήν εδώ πέρα που είναι απλά μια έκθεση μεταφοράς στο κοινοτικό δίκαιο, όπως είπα. Σχόλιο εκτός μικροφών. Δεν, δεν μπορώ εγώ να ανακατευτώ σε ένα ενδοελληνικό πρόβλημα. Κύριο Τούσας. Το θέμα της ενσωμάτωσης της αίτησης στην W στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με άλλα ζητήματα όπως είναι η πειρατεία. Συμφωνώ με την πρότασή σας, με την πρόταση του Πρόεδρου. Και επίσης επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω το εξής. Όλοι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί, οι συνδικαλιστικοί των εργαζομένων στα πλοία, η ITF, η ETF, οι, οι εθνικές ε, συλλογικές ε, συνδικαλιστικές ε, οργανώσεις των αυτεργατών είναι αντίθετη με οποιαδήποτε σκέψη έχει την ενσωμάτωση των αυτεργατών σε όλο αυτό το σχέδιο της στρατηγικοποίησης των πλοίων. Είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα που δεν θέλω να φάω το χρόνο γιατί είναι και άλλο θέμα. Okay, I, I... Ωραία. θα μείνω λοιπόν σε αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Οι ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρήσεων για την ενιαία αγορά πρόκειται πάλι για σχέδιο έκθεσης. Να σας υπενθυμίσω πως η Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς κάνει ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Να μια στιγμούλα για τις 20 κύριες ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρήσεων για την εσωτερική αγορά. Η δε άδειε κυκλοφορία των αυτοκινήτων και τα δικαιώματα των επιβατών είναι τα δικαιώματα τα οποία αφορούν, οι ανησυχίες οι οποίες αφορούν την Επιτροπή μας. Για τα αυτοκίνητα λοιπόν. Η Ένωση έχει εισαγάγει ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης ε, τύπου και καταγραφής για τα οχήματα και έτσι διευκόλυνε την αγορά και μεταφορά αυτοκινήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της αρχής, εάν υπάρχει κοινοτική έγκριση τύπου για ένα αυτοκίνητο και ε, ένα έγγραφο εγγραφής ε, και ασφάλεια μπορεί χωρίς πρόβλημα να εγγράψει το αυτοκίνητο σε άλλο κράτος μέλος. Όμως έχουμε παράπονα από πολίτες που συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες διατυπώσεις που αφορούν ιδιαίτερα την επανακαταγραφή οχήματος σε άλλο κράτος μέλος. Κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Οπότε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ειδικά όταν μιλάμε για την εφαρμογή των σχετικών νόμων στα κράτη-μέλη. Ζήτα επίσης από την Κομισιόν να φέρει ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ε, δοκιμές ε, αξιοπιστίας των αυτοκινήτων για να διευκολύνει την διαδικασία για τα δικαιώματα των επιβατών. Και είχαμε βεβαίως συζήτηση στην έκθεση Taylor και τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μεταφορικά μέσα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι ευθυγραμμισμένος με τα διάφορα πράγματα που γίνονται. Ενιαία εφαρμογή και προστασία των επιβατών σε ολόκληρη την Ένωση έχει σημασία κλειδί για τους πολίτες που ταξιδεύουν και σημαντικό είναι να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείε που κάνουν τις μεταφορές. Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει η νομοθεσία να επικαιροποιηθεί και η Κομισιόν θα πρέπει να δει τα δικαιώματα των επιβατών ε, που ταξιδεύουν με διάφορα μεταφορικά μέσα. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που πρέπει να δούμε. Γι' αυτό τα ζητήματα αεροπορικών επιβατών τα αντιμετώπισε η έκθεση Taylor και ο κύριος Μπαχ θα προετοιμάσει μια έκθεση για τα δικαιώματα των επιβατών σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Είναι σημαντικές λοιπόν αυτές οι εκθέσεις. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω στη γνωμοδότησή μας για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, δεν θέλω ε, εγώ παρά να υπάρχει μια συνέπεια στην προσέγγιση μας. Οπότε βασικά αυτό είναι το θέμα. Ειδικά η εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική για τις ανησυχίες των πολιτών και θέλουν στην Επιτροπή αυτή να κάνουν την έκθεση αυτή. Και ήθελαν να εμπλακούν και άλλες επιτροπές Τα δύο θέματα λοιπόν που μας αφορούν γίνονται στο πλαίσιο της δικής τους έκθεσης. Οπότε η γνωμοδότησή μου δεν αφορά γενικά την εσωτερική αγορά, αλλά αυτούς τους δύο τομείς, γιατί είναι οι δύο τομείς που μας ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Αυτές είναι λοιπόν οι παρατηρήσεις μου και τώρα έχουμε τον κύριο Μπαχ, τον οποίο θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Ως πρόεδρος αναφέρατε τα δύο ζητήματα, αδειοδότηση γιοταχή και δικαιώματα επιβατών. Όσον αφορά την αξιολόγηση γιοταχή σε άλλα κράτη πρέπει να φροντίσουμε πρώτον και το οικονομικό και το διοικητικό κόστος να είναι, ο άχθος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Θα πρέπει δε οι φόροι να αντιμετωπίζονται με ενιαίο κοινοτικό τρόπο, αλλά υπάρχει άλλη μια πτυχή που λέγεται τεχνικός έλεγχος των γεωταχή. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια αμοιβή αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών με βάση κάποιες προϋποθέσεις. Μιλάμε με κοινού ορισμούς, παρόμοιες δοκιμές, μέχρι και ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για μια πανευρωπαϊκή συγκρισιμότητα. Και δυναμική εξέλιξη βεβαίως το περιεχομένου του ελέγχου για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο δική ασφαλεία. Για τα δικαιώματα των επιβατών πράγματι τα τελευταία χρόνια ε, είχαμε μεγάλες πρόοδους για τους επιβάτες στα διάφορα μέσα μεταφοράς και σε αεροπορικές μεταφορές, αλλά όπως αναφέρατε χρειάζεται ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς, ε, όχι μόνο μια κάθετη εναρμόνιση στο κάθε μέσο μεταφοράς αλλά και οριζόντια. Να υπάρχει μια συγκρισιμότητα και καλύτερη πληροφόρηση για να μην έχουμε ακριβώ διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Ιδιαίτερα θεωρώ πως πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα δικαιώματα των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα γιατί όπως διαπιστώσαμε ε, συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να δούμε και τις χρεοκοπίες αεροπορικών εταιριών που συμβαίνουν όλο και συχνότερα και επηρεάζονται εκατομμύρια επιβάτες και εκεί πέρα πρέπει να παραπέμψουμε στο ψήφισμά μας του Νοεμβρίου 2009 και τις προτάσεις που περιέχονται εκεί. Συνολικά θεωρώ πως τα δύο σημαντικότερα ζητήματα τα αναφέρατε ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σάβησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάποιες ε, νέες σκέψεις σε σχέση με αυτά που είπατε εσείς, Πρόεδρε. κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις ή θα μπορούσαμε να θέσουμε και κάποια ερωτήματα ακόμα. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες για τον τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων. Από όσο γνωρίζω όμως, στην πράξη, η τεχνική αυτή ελεγχή είναι πολύ πολύπλοκη. Για παράδειγμα, αν ένα όχημα έχει περάσει από έναν έλεγχο από μία χώρα, δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι εύκολο πάντα να δούμε σε κάποια άλλη χώρα αν το αυτοκίνητο αυτό έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο. Δεύτερη παρατήρηση. Σαφώς είμαστε υπέρ της μείωσης της γραφειοκρατίας. Σαφώς είμαστε υπέρ της απλούστευσης των κανόνων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι παρά όλη αυτή την ενίσχυση των κανόνων Πολλές φορές υπάρχουν αγοραστές που αγοράζουν κλεμμένα αυτοκίνητα, τα οποία μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τους κατάλληλους ελέγχους λοιπόν στα σύνορα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεταφορά ή διακίνηση κλεμμένων αυτοκινήτων. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν επίσης τα ίδια δικαιώματα για όλους τους επιβάτες. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τα πούλμαν και τα λεωφορεία και λυπάμαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε προς αυτό να πετύχει τον αρχικό του στόχο. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα κάποιες μικρές χώρες οι οποίες δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Να σε υπενθυμίσω ότι όταν συζητήσαμε τα δικαιώματα των επιβατών σε λεωφορεία, σε πούλμαν, ακούστηκε τότε μία ιδέα ότι θα έπρεπε δηλαδή τα δικαιώματα όλων των επιβατών για όλα τα μέσα μεταφοράς να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κείμενο. Ακόμα περιμένουν να γίνει κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε με τέσσερις διαφορετικές οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να συγκεράσουμε όλες αυτές τις οδηγίες σε ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστα. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας, για την έκθεσή σας. Έχετε αναλάβει αρκετές εκθέσεις. Στο θέμα των αυτοκινήτων, συμφωνώ 100%. Εάν αγοράσετε ένα αυτοκίνητο στο Βέλιο στη Γαλλία, έχουν άδεια αυτά τα αυτοκίνητα. Υπάρχει και η άδεια από τον κατασκευαστή. Δεν έχει σημασία αν μεταβαίνει ε, κανείς αν ε, πηγαίνει από μία χώρα σε άλλη. Δεν ήξερα ε, για τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Έχει δίκιο ο συνάδελφος και βεβαίως μπορεί κανείς ε, να μεταβεί από μία χώρα στην άλλη γιατί το Σέγγεν δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και σύνορα τα οποία δεν μπορούν να παραβιαστούν. Υπάρχει ένα θέμα, αλλά θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία ως προς τα δικαιώματα των πιβατών, Ο Μάλκομ είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος. Ε, δέχομαι ότι η ΙΜΚΟ έχει πολλή δουλειά, αλλά δεν ξέρω πώς ε, κατέληξε έτσι. Δηλαδή ασχοληθήκαμε με τα δικαιώματα επιβατών εδώ και χρόνια και επαναλαμβάνουμε τα ίδια χρόνια και χρόνια. Δεν λέω ότι υπάρχουν ε, κακές προθέσεις, αλλά υπάρχουν πολλές επικαλύψεις. Εμείς ε, έχουμε τον κύριο λόγο και δεν νομίζω πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. ως προς τη πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για την δοκιμή των αυτοκίνητων χρειάζεται πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Ίσως αυτό μπορείτε να μου το αποσαφηνίσετε. Με συγχωρείτε που περνάω από το ένα θέμα στο άλλο. Μίλησα για τα δικαιώματα των επιβατών. Έχουμε κανονισμούς, οδηγίες για τα δικαιώματα των επιβατών. Γιατί πρέπει να τα υποβάλουμε όλα στον ίδιο κανονισμό, γιατί να τα, να τα τάσουμε κάτω από τον ίδιο κανονισμό. Υπάρχουν ε, διατροπικές μεταφορές, υπάρχει διαφορά, δεν πρόκειται για μια κοινή θεματική. Εάν πρόκειται κανείς να χρησιμοποιεί πλοίο ή όχημα, δεν καταλαβαίνω γιατί το τονίζουμε, γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, ας ε, μην φτάσουμε σε σημείο κορεσμού. Καλά τα καταφέρνουμε το τομέα μεταφορών, ας μην ε, ε, επαναλαμβανόμαστε γιατί αποδυναμώνουμε το κείμενό μας. Σας συγχαίρω για την εργασία σας, όπως συνήθως, και σας εύχομαι καλή έκβαση. Δεν έχουμε κανέναν από την Επιτροπή, διότι δεν αφορά μεταφορές, αλλά περισσότερο εσωτερική αγορά. Αυτό θα έβαζε η τα δικαιώματα των επιβατών, άρα δεν μπορούσαμε να το αγνοήσουμε. Έχετε δίκιο. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Μπάξ και ο Γιώργος έχει αναλάβει και ένα άλλο θέμα για το cross-modal Έχετε δίκιο. Καλύτερα να έχουμε ένα ε, νομοθετικό όχημα και όχι πολλά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται με την έκθεση του κυρίου Μπαξ. Κυρία Φώστερ, ως προς το δεύτερο θέμα, ως προς την αξιοπιστία των οχημάτων, στην Ευρώπη υπάρχουν 27 διαφορετικά πρότυπα Άρα όταν κανείς μεταβαίνει από μια χώρα σε άλλη και πρέπει να ξανακαταγράψει το όχημα, πολλές φορές θα πρέπει να προηγηθεί ο τεχνικός έλεγχος Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας ενίος τεχνικός έλεγχος ως προς την αξιοπιστία των οχημάτων για να διευκολύνει την ε, ένταξη, την καταγραφή σε άλλο κράτος μέλος. Λοιπόν, 8 Μαρτίου, προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών, ψηφίζουμε στις 24 Απριλίου, 19 Ιουνίου, στη συνέχεια η ΙΜΚΟ θα ψηφίσει στις 19 Ιουνίου. 8 Μαρτίου. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Τώρα περιμένουμε την κυρία Τσικάου για την έκθεσή της. Okay, I'm told we may need to break. I'd rather... Ίσως πρέπει να διακόψουμε. Να προσπαθήσουμε να έρθει κάπως νωρίτερα από τις 11 η κυρία Τσικάου, αν γίνεται γιατί είναι πολύ σημαντική η έκθεση της για τους ε, ταχογράφους. Λοιπόν, διακοπή 10 λεπτών μέχρι να βρούμε την κυρία Τσικάου. 10 Okay, I'm την κυρία Τσικάου να έρθει εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και θα περάσουμε όταν έρθει στην εξέταση της έκθεσης για τους ταχογράφους. Um, before, just to give Sylvia a minute to Πρωτού πάρει το λόγο η Σίλβια, να σας δώσω και το χρονοδιάγραμμα. Αρχικά η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν η 6η Μαρτίου και την επεκτείναμε μέχρι την 15η Μαρτίου. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι πλέον η 15η Μαρτίου 12 το μεσημέρι και ελπίζουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Απρίλιο. Η αλλαγή ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών πέρασε από την 6η στη 15η Μαρτίου. Αυτά. Ψηφιακή ταχογράφη. Αυτό είναι το επόμενο μας θέμα. Δίνω το λόγο στην κυρία Τσικάου. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία ιδιαίτερα την Ελβίρα για τη συνεργασία και για τον τρόπο που συνεργαστήκαμε. Επίσης όλους τους σκιώδεις θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί συνεργαστήκαμε άριστα και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Το θέμα αυτό είναι άκρος ενδιαφέρον, είναι τεχνικής υφής, άκρος ενδιαφέρον και έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με την τήρηση της ε, νομοθεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Δεν θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το ιστορικό της εισαγωγής των ταχογράφων. Θα ήθελα να σας πω μόνο ότι αρχίζοντας από το 85 Είχαμε τους αναλογικούς ταχογράφους που ακόμα χρησιμοποιούν ορισμένα οχήματα που ε, κυκλοφόρησαν πριν από την 1η Μαΐου 2006. Μετά από την 1η Μαΐου του 2006 υπάρχει η πρώτη γενεά των ψηφιακών ταχογράφων, όμως υπάρχουν προβλήματα διότι καταπατάται η κοινωνική νομοθεσία δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος ανάπαυσης και η μέγιστη περίοδος οδήγησης. Δυστυχώς κουράζονται ιδιαίτερα οι οδικοί και αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κυκλοφορία. Επίσης οι μεγάλες εταιρείες δεν τηρούν την κοινωνική νομοθεσία για να έχουν ένα ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να μειώσουν τις τιμές. Γιατί ε, η πληρωμή των οδηγών αποτελεί το 30-50% του συνολικού κόστους. Οι ταχογράφοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί ακόμα σήμερα όσο θα έπρεπε. Εισήχθη για την καταγραφή και μόνο και δεν ερμηνεύει σωστά, δεν αντικατοπτρίζει την κοινωνική νομοθεσία. Γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της Κομισιόν, διότι προβάλλει διευκρινήσεις στο κείμενο και βελτιώσεις ως προς την λειτουργία του ψηφιακού ταχογράφου. Θέλουμε την επικαιροποίηση του κειμένου για να μην υπάρχουν, να μην γίνονται απάτες, να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο και να τηρηθεί η κοινωνική νομοθεσία. Θα θέλαμε επίσης να έχουμε επέκταση της χρήσης των ψηφιακών ταχογράφων και να εισαχθούν οι ευφυείς ταχογράφοι έτσι ώστε να υπάρχει επικοινωνία τηλεεπικοινωνία και έλεγχος. Επίσης να γίνεται εισαγωγή της ε, αυτόματη καταγραφή της, ε, καταγραφή της ακριβούς θέσης με το σύστημα GNSS. Επίσης να έχουμε συγχώνευση λειτουργικών δυνατοτήτων της κάρτας οδηγού με την άδεια οδήγησης και εδώ θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι θα πρέπει να εισηχθεί και ένα σωστό νομικό πλαίσιο για την έγκριση συνεργείων και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, ένας ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης των κυρώσεων, Επίσης, ως πέμπτο, υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση στους ελεγκτές και έκτον, μέτρα εξαίρεσης ορισμένων οχημάτων από την υποχρέωση χρήσης ταχογράφου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι δεν έχουμε εισαγάγει παρά μερικές και μόνον αλλαγές, οι οποίες δεν επαρκούν για την εισαγωγή των ταχογράφων νέας γενεάς και γι' αυτό έχουμε εισαγάγει και ορισμένες τροπολογίες. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν αυτό το ελεγκτικό υλικό υποδομής έτσι ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν η ταχογράφοι νέας γενεάς, ψηφιακή ταχογράφοι νέας γενεάς, για να μειωθούν και οι έλεγχοι και να υπάρχει τηλεεπικοινωνία και τηλεέλεγχος. Δηλαδή ο ψηφιακός ταχογράφος νέας γενεάς ενέχει και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ποιήσεις όταν σταματάει το όχημα για έλεγχο έτσι ώστε να μην χάνεται χρόνος σε ορισμένες διενέργειες ελέγχου. Δηλαδή να μην το σταματάνε το όχημα συνέχεια για ελέγχους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό το μέσον ελέγχου και οι ελεγκτές να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, διότι πολλές φορές, και το συζήτησα με την ε, Πολ, δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση. Μας είπε λοιπόν ο φορέας αυτός ότι δυστυχώς στα κράτη-μέλη οι έλεγχοι διενεργούνται κατά διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό γίνονται και καταστρατηγήσεις της ε, κοινωνικής νομοθεσίας. Επίσης, έχουμε εισαγάγει νέε ε, διατάξεις για την προστασία δεδομένων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Και λαμβάνουμε υπόψη και την εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Προτείναμε και μάλλον διαπιστώσαμε ότι στα διάφορα νομοθετικά πλαίσια γίνεται χειραγώγηση των ε, ταχογράφων και αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο έγγραφο ελέγχου και του ταχογράφου και αυτό το ορίζουμε μέσω τροπολογίας. Έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή ταξινόμηση των ε, καταστρατηγήσεων έτσι ώστε όταν κανένας πειράζει τον ταχογράφο και μετατρέπει τα δεδομένα οι κυρώσεις να είναι πολύ αυστηρές το πλαίσιο κυρώσεων να είναι πολύ αυστηρό. Για να μην ε, μπορεί κανείς να προβαίνει σε σε παρόμοια εγχειρήματα, να μην πειράζει τους ε, ταχογράφους και να αλλάζει τα δεδομένα. Ζητήσαμε την εντατικοποίηση των ελέγχων, γιατί φαίνεται πολλές φορές και από τα εργοστάσια γίνεται πολλές φορές αυτή η μετατροπή των ταχογράφων. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και τις δραστηριότητες, τι γίνεται ακριβώς σε επίπεδο κατασκευής. Στις κατεξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται το Συμβούλιο ζήτησε να λάβουμε υπόψη και τις εκτελεστικές ε, πράξεις, αλλά εμεί δεν έχουμε ρόλο στις εκτελεστικές πράξεις, μόνο στις κατεξουσιοδότηση. Και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στις κατεξουσιοδότηση αποκλειστικά. Σε σχέση με την άδεια, τις άδειες οδήγησης και το ενιαίο έγγραφο, μπορούμε να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο που να αφορά και τις άδειες οδήγησης, ανάλογα με τις επαγγελματικές κατηγορίες και να μιλάμε για ένα ενιαίο έγγραφο για να αλλάξουμε και την οδηγία που αφορά τις άδειε οδήγησης. Προσωπικά πιστεύω ότι από τεχνικής πλευράς θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το πλαίσιο ενιαίου εγγράφου είναι εφικτό. Αλλά σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν δύο υπεύθυνοι. Το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πλαίσιο της ενιαίας, ε, της άδειας οδήγησης και του ενιαίου αυτού εγγράφου μεταφορών. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτά τα δύο έγγραφα σε ένα. Υπάρχουν δύο συστήματα μηχανογράφησης, αλλά μπορούν να πλαισιωθούν ενιαία. Όταν μιλάμε για άδεια οδήγησης και για επαγγελματικές, επαγγελματική άδεια, θα πρέπει να έχουμε μία ευφύη κάρτα και μία ευφύη κάρτα επίσης και για τον ταχογράφο. Δεν είμαι πεπισμένη όμως ότι η παρούσα πρόταση της Επιτροπής είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι το καταλληλότερο μέσο. Και αυτό το λέω διότι από την, ε, τα έγγραφα που είδα, από την τεκμηρίωση, βλέπω ότι η άδεια οδήγησης είναι πολύ πιο ασφαλής από ότι το, το καρνέ του οδηγού. Και τη στιγμή που θα έχουμε μία και μόνο ευφυή κάρτα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά και ασφαλής. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα δύο έγγραφα τα οποία θα αποτελέσουν ένα, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς εισαγάγονται όλα τα δεδομένα που αφορούν τα επαγγελματικά δεδομένα και τα επαγγελματικά εχέγγυα. Πιστεύω στην ενιαία κάρτα, αλλά θα πρέπει να διενεργηθεί μια μελέτη αντικτύπου για να δούμε ποιο είναι και το εμπλεκόμενο κόστος για τα κράτη-μέλη σε σχέση με τα δύο αυτά συστήματα που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη και να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς. Θα πρέπει λοιπόν να διενεργηθεί μία μελέτη αντικτύπου έτσι ώστε να μειωθεί και η αντίσταση των κρατών μελών για την ενιαία αυτή πλαισίωση. Γι' αυτό θα υποβάλουμε και ορισμένες τροπολογίες στο σχετικό άρθρο για την ενιαία πλαισίωση για να ζητήσουμε τη διενέργεια μελέτης αντικτύπου και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να προβάλλει μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Υπάρχουν όμως ορισμένες ενδείξεις ήδη για την ενσωμάτωση αυτών των δύο εγγράφων και επιστοποιήσεων. Θα σταματήσω εδώ. Περιμένω τις απόψεις σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μας απασχολεί όλους και υπάρχει και πολύ ισχυρός αντίκτυπος στις οδικές μεταφορές. Γι' αυτό πρόθεσή μας είναι να έχουμε μια καλή έκθεση, έναν καλό κανονισμό που να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και από τις επιχειρήσεις και από τους ε, οδηγούς και από τις ελεγκτικές αρχές. Και ελπίζω με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το οποίο να είναι χρήσιμο για τον τομέα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mrs. for your remarks and your report. Now for the PPE. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Higgins από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κυρία Τσικάου για αυτά τα οποία έκανε. Συναντηθήκαμε, συζήτησε λεπτόμερος με τους σκιοδησηγητές και συμπεριέλαβε πολλές ε, σκέψεις μας. Είναι τεχνικό το ζήτημα όπως είπε και πρέπει να φροντίσουμε να είναι σωστό. Σε σχέση με το άρθρο 19 παράγραφος 4 λέει τα κράτη-μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγουν ε, συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ συνεργείων ε, και μεταφορικών εταιριών. Συγκεκριμένα, αν μια μεταφορική εταιρεία ε, είναι εγκεκριμένο συνεργείο, δεν θα επιτρέψει να εγκαταστήσει και να βαθμονομήσει το σύστημα στα οχήματά της. Νομίζω, τώρα όταν μιλάμε για αξιόπιστες εταιρείε όπως η DHL και η UPS, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και εγκατάσταση και ε, επιθεωρήσεις γιατί είναι αξιοσέβαστες εταιρείε. Βεβαίω πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ε, να υπάρχει κανένας κανένα λαμόγιο, αλλά θα πρέπει ε, νομίζω και να ελέγχονται και αυτοί από καιρού καιρών αλλά να έχουν τη δυνατότητα να βάζουν τα συστήματα αυτά και να τα συντηρούν την ίδια τη συσκευή για την ε, τροπολογία 57 κάπου πρέπει να τονίσουμε πως ταχογραφή είναι ένα από τα συστήματα για την οδική ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει μια βάση δεδομένων πανευρωπαϊκή των μεταφορικών εταιριών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και συνδέεται με την τροχέα. Και η τροχέα μπορεί να δει το φορτηγό και να δει τι έχει γίνει στις προηγούμενες επιθεωρήσεις. Το πρόβλημα, ο κίνδυνος είναι ό,τι και αν κάνουμε πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα μπορέσουν να παρακάμψουν τη συσκευή και να εξαπατήσουν το σύστημα. Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση της κυρίας Τσικάου να ενσωματωθεί η κάρτα του ταχογράφου με το δίπλωμα του οδηγού γιατί είναι κομμάτι του ίδιου πράγματος. Τροπολογία 37. Τώρα. Αυτή έχει προελθεί από τα παραρτήματα και έχει μπει κατευθείαν στο διατακτικό. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί πρέπει να ορίσουμε ξεκαθαρά τι ορισμούς έχουμε σε σχέση με το τι ακριβώς είναι ταχογράφος. Η τροπολογία 45 συμφωνώ. Θεωρώ πως η πρόταση της Κομισιόν είναι φευρή η κυρία Τσουκάου προτείνει δύο χρόνια. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να μην λειτουργήσει σε δύο χρόνια. Αν υπάρχει η συσκευή, ας γίνει. Για δική ασφάλεια μιλάμε. Τροπολογίες 91 και 95. Και πάλι επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Τσικάου για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Δεν έχει νόημα να επενδύσουν οι εταιρείε και η αστυνομία. Είναι αστυνομικοί, δεν μπορούν να βρουν τυχόν απάτη και είναι περίπλοκο το ζήτημα. Είναι τεχνικό επίσης και δεν επαρκεί να μην ε, ορίσουμε ε, το ποια είναι η εκπαίδευση των αστυνομικών. Πρέπει να υπάρχει στην εκθέση και τέλος για την τροπολογία 81 αυξημένη έλεγχη των συνεργείων. Το ορίζω, Λέει να αυξηθούν οι έλεγχοι από το 10% που είναι η πρόταση κομισιόν στο 20% όλων των, των συνεργείων. Καλύτερα να γίνονται επιθεωρήσεις τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, όχι κάθε δύο χρόνια. Αυτό προτείνω. Και καλωσορίζω την εκθέση σας. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ για του φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω πως ο κύριος Higgins βεβαίως είναι Ιρλανδός. Ναι, ναι, δεν ήξερα τελικά, δεν ήμουν σίγουρη αν ήσασταν από τη Μεγάλη Βρετανία ή την Ιρλανδία. Σας ζητώ συγγνώμη. Πάντως μιλάτε αγγλικά. Συμφωνώ λοιπόν με τον Ιρλανδό συνάδελφο κύριο Χίγκινς απολύτως και να ευχαριστήσω την κυρία Τσικάου για την πολύ καλή αυτή έκθεση, για την όλη εργασία που έκανε και στο παρελθόν μας κάλεσε μας τους Κιώδης πάρα πολλές φορές και συζητήσαμε εκτενώς όλα τα ζητήματα, όλες τις ανησυχίες που είχαμε για την πρόταση αυτή και μιλήσαμε διεξοδικά για το τι θα πρέπει να καλύπτει η έκθεση αυτή. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτή τη μέθοδο εργασία. Μ' αρέσουν επίση και οι τροπολογίε όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Διευκρινίζουν αρχικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέγεται ότι θα πρέπει να επεξεργάζονται, να είμαστε σε θέση να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του τεχογράφου, προστατεύοντας όμως τα προσωπικά δεδομένα των οδηγών. Υπάρχουν όμως κάποιες ασάφειες. Ίσως θα πρέπει να γίνει και μια σχετική τροπολογία. Για παράδειγμα, τι είναι τα απαραίτητα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι εδώ. Η πρόταση του ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν το GNSS είναι καλή. Τι θα γίνει όμως για, τα, για τις επιπρόσθετες δαπάνες της εγκατάστασης της αντένας του δέκτη και το καθεξής μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της δαπάνης εγκατάστασης του ταχογράφου και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Κάτι που δεν μου αρέσει όμως καθόλου είναι οι εξαιρέσει που προβλέπονται ε, στην δική σας την τροπολογία την υπαριθμών 2, η οποία αντιτίθεται ουσιαστικά στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν αναφερθήκατε καθόλου στις προτινόμενες εξαιρέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιορίζουν ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα τον τομέα του εμπορίου ή της ε, εταιρείας logistics. Και νομίζω ότι το 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν τότε έτοιμη να προχωρήσει από τα 15 στα 150 χιλιόμετρα. Είχε συζητήσει για το ζήτημα αυτό με τα κράτη-μέλη. Και Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό ιδίω για τους μη επαγγελματίε οδηγού και θα ήθελα λοιπόν ως προς αυτό να κάνω μια τροποποίηση, μια τροπολογία για τη θέση σε ισχύ του κανονισμού που σχετίζεται και με το GNNS από 48 σε 24 μήνες. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί ξέρετε ότι η νέα τεχνολογία θα πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί και θα πρέπει να γίνει και μια εκπαίδευση, μια κατάρτιση του προσωπικού. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Τώρα η συχνότητα των ελέγχων και αναθεώρηση των ταχογράφων αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Χίγκινς, Λέτε τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε μια ενημερωμένη, επικαιροποιημένη τεχνολογία, ενδεχομένως όμως η διαδικασία να είναι κάπως γραφειοκρατική και όχι απαραίτητα τόσο αναγκαία. Προτείνεται επίσης και μία ομοιόμορφη άδεια πιστοποίηση για τους ελεγκτές, ότι θα πρέπει να πιστοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο οι ελεγκτές αυτοί. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και δίνεται έτσι και η δυνατότητα να χρησιμοποιούν την απαραίτητη πιστοποίηση και την απαραίτητη υποδομή αυτοί οι ελεγκτές. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την πρόταση. Έχετε συμπεριλάβει μία δεσμευτική κατηγοριοποίηση κάποιων πολύ σημαντικών παραβιάσεων προκειμένου υπάρχει ένα, θετικό, ένα θεμητό πεδίο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, αλλά αυτό περιορίζει κάπως την ευελιξία των κρατών μελών να μπορούν να κάνουν αυτά τη δική τους συναξιολόγηση. Γι' αυτό το λόγο θα υποβάλω και μια τροπολογία. Προσθέσετε κάποιες βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση, τη χρήση, τον έλεγχο, τη δοκιμή των ταχογράφων και για τη λειτουργία των ταχογράφων, τα δεδομένα που θα πρέπει να καταγραφούν, την πρόσβαση στα δεδομένα, την προστασία των δεδομένων αυτών και όπως είπα στην αρχή εν γέννη μ' αρέσει η έκθεσή σας και απλώς θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Εν γέννη πάντως πιστεύω ότι έχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, ναι. ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσικάου πολύ καλή έκθεση. Έχουμε προβλήματα γιατί τι γίνεται. Ε, μειώνονται συνεχώς οι συνθήκες εργασίας των οδηγών διεθνών μεταφορών και αυτό είναι λυπηρό για την οδική ασφάλεια. Κάποια πράγματα που θα ήθελα να παρατηρήσω επιπροσθέτως. Μεγάλο πρόβλημα είναι ο χρόνος και οι εγκαταστάσεις ανάγνωσης για το κατέβασμα των ψηφιακών αυτών δεδομένων. Χρειάζεται τόσο χρόνος που αποτελεί πρόβλημα. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Θεωρώ επίσης πως μια... πρέπει να υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή που θα δίνει τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στους οδηγούς γιατί η πίεση εδώ πέρα στον οδηγό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτές είναι πληροφορίες που μου είπαν και οι αρχές. Δηλαδή οι οδηγοί έχουν δυσκολίες. Γιατί ε, βεβαίω αντιμετωπίζουν κινδύνους με τη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει πως αν ε, παίζεται ένα παιχνίδι στις πλάτες ε, του οδηγού, δεν σημαίνει πως ε, μπορούμε έτσι απλά να βελτιώσουμε την κατάσταση για τον ίδιο τον οδηγό. Εκεί πέρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Βεβαίω υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν για λογαριασμό τους, αλλά οι περισσότερες παραβιάσεις δεν οφείλονται στους οδηγούς, αλλά στις εταιρείε που τους απασχολούν. Θεωρώ και αυτό φάνηκε στην τελευταία περίοδο και η δική μας δυσκολία είναι πως τα δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη δεν είναι πλήρη. Υπήρξε η προσπάθεια να γίνει μία μελέτη για αυτό το θέμα για το πώς ε, είναι χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης, ε, τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος και εκεί πέρα αποδείχτηκε, νομίζω δεν ξέρω 2007 ή 2008, πως τα τελευταία αξιόπιστα δεδομένα ήταν το 2001. Ήδη δηλαδή δεν έχουμε καν δεδομένα να βασιστούμε. Και να σας υπενθυμίσω ο τότε επίτροπος μας υποσχέθηκε πως θα ασχοληθεί με την επιβολή στα κράτη-μέλη. Γιατί έχουμε πρόβλημα, ειδικά όσον αφορά τους ψηφιακούς ταχογράφους. Και την επιτήρηση. Εάν δεν έχουμε δεδομένα από τα κράτη-μέλη που να είναι αξιόπιστα και πρόσφατα, τι δύσκολο να, μπορέσουμε, να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Γιατί είναι τεχνικός ο τομέα και ξέρετε, η εφευρετικότητα στην παραβίαση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε πρέπει και τα κράτη-μέλη να ε, φροντίσουν να έχουν πληροφορίες και να δίνουν στην Κομισιόν πληροφορίες πρόσφατες για να αντιδρά και η Κομισιόν εγκαίρως. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Και πάει όλη η στρατηγική χαμένη. Γιατί εμείς βγάζουμε εδώ πέρα ωραίους φιλόδοξους νόμους και κάποια κράτη-μέλη λένε δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Δηλαδή η πυκνότητα των ελέγχων διαφέρει πάρα πολύ και γίνεται επιλεκτικά τα πράγματα. Εμείς χρειαζόμαστε λοιπόν και να δούμε πού γίνεται η παραβίαση αυτών των μηχανημάτων και θα πρέπει και μέσω της Κομισιόν να προειδοποιηθούν τα κράτη-μέλη, να δίνουν πρόσφατα δεδομένα στην Κομισιόν. Επίσης, Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Στην όλη διαχείριση αυτών των μηχανημάτων. Π.χ. αν σβήνει κάποιος το φορτηγό και μετά δεν υπολογίζεται κάτι τέτοιο ε, ως χρόνος εργασίας Αυτό το οποίο μας λένε δηλαδή και οδηγεί. Κάτι πρέπει να, να κάνουμε. Τέλος για τις πράξεις κατεξιοδότηση. Είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τις ορίσουμε σωστά και να περιορίσουμε το τι επιτρέπεται να κάνει η Κομισιόν και να αλλάξει. Γιατί για να μπορεί να αντιδράσει γρήγορα. Από την άλλη, δεν θέλω να δώσουμε μια αξιοδότηση στην Κομισιόν να κάνει ό,τι θέλει. Δεν την εμπιστεύομαι και τόσο. Γιατί αν δούμε πώς γίνεται η εφαρμογή στα κράτη-μέλη, φαίνεται πως δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε εμείς εδώ μέσα. Γι' αυτό, ναι, σε πράξεις κατεξιοδότηση, αν είναι όμως ακριβώς ορισμένες, γιατί έτσι οι γενικές εξουσιοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια δεν απέδωσαν, παλαιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα, τέλος πάντων. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να ε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για εμένα, για τη μεταφορά των ζώων θα πρέπει να περάσουμε στους ψηφιακούς ταγωγράφους για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ειδικά στη μεταφορά των ζώων, τα κόλπα εκεί πέρα που γίνονται με τα δικαιώματα των ζώων και των εργαζομένων είναι μεγάλα. Το πρόβλημα παραμένει σχέση μεταξύ α, ώρας εργασίας του οδηγού και ώρας ανάπαυσης. Τα έχουμε συζητήσει. Είναι ανοιχτό το ζήτημα. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την ε, πλήρη αυτή εισαγωγή που έκανε στην εκθεσή της. Νομίζω ότι αναμφίβολα εξελίσσεται η τεχνολογία πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να την εκμεταλλευτούμε. Και πρέπει να δούμε βέβαια πώς έχει εξελιχθεί ο ταχογράφος και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που επινοήθηκαν ποτέ, τουλάχιστον για την ασφάλεια και καθώς εξελίσσεται και η τεχνολογία, καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες άλλες υπηρεσίε, όπως ο γεωγραφικός εντοπισμός και κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται πολύ περισσότερο και το ίδιο το επίπεδο της ασφάλειας. Τώρα για τη συγκεκριμένη έκθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτόν τον δρόμο. Έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκθεση της κυρίας ΤικάΟ. Και από ό,τι φαίνεται πολλά παραρτήματα έχουν περάσει τώρα στα άρθρα, και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί όταν έχουμε παραρτήματα για τεχνικές εκθέσεις, τα παραρτήματα πολλές φορές μπορούν να εξελιχθούν εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε από την νομοθετική διαδικασία του Κοινοβουλίου. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει κανείς όταν περνάει τα πάντα στο διατακτικό ενός νομοθετικού κειμένου. Επομένως, έχω μια κάποια ανησυχία όσον αφορά το περιεχόμενο των άρθρων, όπου ουσιαστικά έχουμε ενσωματώσει το περιεχόμενο από πάρα πολλά παραρτήματα. Αυτό μου προκαλεί μια κάποια ανησυχία. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε σαφώς στο μεγάλο βαθμό απάτης. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν είναι ε, ειλικρινείς, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι όλος ο τομέας των ε, μεταφορών, ότι όλοι οι οδηγοί παντού στην Ευρώπη είναι μικροαπατεώνες και προσπαθούν να βγάλουν χρήματα παραβιάζοντας τον ταχογράφο. Δεν είναι δίκαιο να πούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως σαφώς κάποιοι άνθρωποι, ένα ποσοστό οδηγών, που προσπαθούν πολλές φορές, ιδίως με την παλαιότερη τεχνολογία ταχογράφων, να παρακάμψουν του ταχογράφους αυτούς. Πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση που κάνουμε, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα ασχολούμαστε με έναν μικρό στόλο οδηγών. Επομένω επομένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και, ο, και ο περαιτέρω εξοπλισμός που να χρειαστούν να έχουν στο μέλλον δυο τρει παρατηρήσει τώρα πιο συγκεκριμένε. Όσον αφορά τα εγκεκριμένα συνεργεία για τον ταχογράφο που θα πρέπει να, εγκαταθ... να εγκαταστούν από τους κατογράφους, διαφωνώ με αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση των κρατών μελών, ενδεχομένω να είναι δύσκολο για κάποια κράτη-μέλη. Ο κύριο Χίγκιν αναφέρθηκε σε αυτό. Στο δικό μου το κράτο. έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα, το κατάλληλο σύστημα που λειτουργεί εδώ πέρα και πάρα πολλές δεκαετίες και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την εγκατάσταση των ταχογράφων αυτών θα μπορούσαν ποτέ να προχωρήσουν σε απάτη. Έχουν ε, κάποιες επιχειρήσεις λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να διατηρήσουν ε, την δραστηριότητά τους αυτή και όχι να τη χάσουν εξαιτία μιας κοινοτική νομοθεσίας ε, η οποία θέλει να διοργανώσει το σύστημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένω, δεν θέλουμε να γίνει μια εξολοκλήρου αλλαγή στο υφιστάμενο σύστημα. Προφανώ θα πρέπει να δούμε και τη συχνότητα των ελέγχων, προκειμένου τα συνεργεία αυτά να λειτουργούν σωστά. Συμφωνώ με αυτό. Κάποιε άλλε παρατηρήσει τώρα όσον αφορά την συγχώνευση. Ενδεχομένω να πρέπει να συγχωνευτεί, να ήταν ιδανικό να συγχωνευτεί ο ταχογράφο με την άδεια οδήγηση. Στην πράξη δεν νομίζω θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα και ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να μην θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί ε, η συγχώνευση αυτή στην πράξη θα μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν σε αυτό. Θα πρέπει απλώς ε, οι οδηγοί να έχουν την απαραίτητη άδεια και οι ταχογράφοι να είναι επιστοποιημένοι και να λειτουργούν σωστά. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλε άδειε. Μια τελευταία παρατήρηση από συνάδελφών που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, για τους οδηγούς από τρίτες χώρες. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλούς οδηγούς στην Ευρώπη, πλέον από την Ουκρανία ή από τη Ρωσία και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι οδηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν ε, πάρα πολλά κριτήρια. Ποια είναι η απόψη όμως της ηγήτριας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους οδηγούς από τρίτες χώρες όπως η Ουκρανία ή η Ρωσία. Δεν λέω απαραίτητα ότι είναι ύποπτοι, αλλά τι κάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Θα έχουν όλοι αυτοί τους ίδιους ψηφιακούς ταχογράφους. Και τελευταία παρατήρηση. τι κάνουμε με τις ε, υπηρεσίες επιβολής της νομοθεσίας από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ξέρετε ότι ε, αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να συμμορφώνονται, για παράδειγμα, τα φορτηγά με του κανόνε που ισχύουν σε κάθε κράτο μέλο. Οι κανόνε μα αυτοί διαφέρουν από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Σαφώ θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση για το ζήτημα αυτό, για του ελέγχου αυτού σε κάθε κράτο μέλο. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να μα απασχολήσει λίγο περισσότερο το ζήτημα αυτό. Είναι αρκετά πολύπλοκο και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εισηγήτρια για την εργασία που έχει κάνει σε αυτό τον τομέα. Σα ευχαριστώ. Θέλετε το λόγο, γιατί δεν μας είπατε αν θέλετε να μιλήσετε από την ομάδα σας. Mm, ναι. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, δεν έχω καμία παρατήρηση. Mr. Yeah, Κύριε Σερτού, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω την κυρία Τσικάου για τη δουλειά που έκανε. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Και έχω και μια παράκληση. Είναι σημαντικό αυτά τα οποία έκανε η συγκήτρια να τα διευκρινίσουμε. Δεύτερον, και εδώ πέρα θέλω να σας υποστηρίξω πως και η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν πρέπει να μειωθεί. Δηλαδή, όταν μεταδίδονται τα δεδομένα αυτά, πρέπει να προστατεύονται. Αλλά, κάτι άλλο. Έχω μια παράκληση. Σήμερα, κατά βάση, μιλάμε για οδήγηση και για ανθρώπους που ασχολούνται με τις οδικές μεταφορές. Ότι πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις οι υποχρεωτικές δεν το συζητάμε. Θέλω να εστιάσω την προσοχή σας σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά αλλά πρέπει να οδηγήσουν για να πάνε να κάνουν την κανονική τους δουλειά. Μιλάμε για διάφορους τεχνίτες και μάστορες κτλ. και υπάρχει ο λεγόμενος κανόνας ε, των 50 χιλιόμετρων ακτίνας νομίζω δράσης και η Κομισιόν εάν δεν κάνω λάθος θέλει να επεκτείνει τον κύκλο αυτό από τα 50 στα 100 χιλιόμετρα καλό είναι αυτό χωρίς βεβαίως να μειώνεται η προστασία των εργαζομένων θεωρώ όμως πως θα πρέπει να σκεφτούμε τις ε, περιοχές της Υπέθρου. Στην Υπέθρο οι επιχειρήσεις είναι κυρίως μικρομεσαίες. Και εκεί πέρα αυτές είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και οι περιοχές αυτές έχουν το πρόβλημα πως ακριβώς οι διάφορες βιοτεχνίες και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να οδηγήσουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε να ξεκινήσουν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω. Ε, ε τα κλασικά, ε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπογιατζίδες, ε, άνθρωποι που φτιάχνουν στέγες και τα λοιπά. Και συχνά πάνε, ξέρω φανταστείτε ας πούμε τα δάση της Βαβαρίες, ε, οπουδήποτε Μόναχο, Νιρεμβέργη και πολύ γρήγορα ξεπερνάνε αυτό το όριο των 50 χιλιόμετρων και των 100 ακόμα. Και θέλω να παρακαλέσω το όριο αυτό να επεκταθεί ακριβώς για να μην έχουν ε, μειονέκτημα οι μικρές αυτές περί επιχειρήσεις. Εγώ θα προτιμούσα τα 200 χιλιόμετρα, αλλά αν δεν γίνεται τουλάχιστον 150 για να βοηθήσουμε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις ε, που δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί, οδηγούν για να πάνε να κάνουν την δουλειά τους. Χωρίς όπως είπα να μειώνεται η προστασία των οδηγών. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να με στηρίξετε σε αυτό. Ευχαριστώ. Σκόχ. Ευχαριστώ την κυρία Τσικάου για την πολύ καλή της έκθεση. Κυρία Τσικάου, ε, μιλήσατε για το πόσο ο ψηφιακό ταχογράφο θα βοηθήσει το ωράριο, τι κοινωνικέ διατάξει. Πρέπει να είναι απλό και αποτελεσματικό το σύστημα και κυρίω βέβαια να βελτιώσει την οδική ασφάλεια. Ο ψηφιακό ταχογράφο δεν ισχύει για τα γιοταχή. Επί τη αρχή σωστό είναι αυτό και το χαιρετίζω. Αν και καμιά φορά ανησυχώ ε, για το όταν ε, κανείς ε, και, και εγώ ακόμα μετά από μια εβδομάδα εργασίας οδηγώ και επιστρέφω στην πατρίδα μου αλλά συμφωνούμε πως όταν μιλάμε για πυροσβεστικά οχήματα, στενοφόρα κτλ προφανώς πρέπει να εξαιρεθούν αλλά και για μικροβιοτέχνες που δεν είναι ο βασικός τους στόχος και η δουλειά η οδήγηση απλά οδηγάνε για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, μια υπηρεσία την οποία παρέχουν και θα πρέπει άρα να εγγυηθούμε, συμφωνώ εδώ πέρα με τον συνάδελφο, έναν επαρκή κύκλο ε, για να μπορούν αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Κύριο Σπέρκερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας συγχαίρω για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα τέσσερα σημεία να αναφέρω. Πρώτον, το ανέφεραν προλαλήσαντες. Αναφέρεται στην τροπολογία 2 που μιλάμε για τις εξαιρέσεις. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θεωρώ πως είναι σαφές και αιτιολογημένο και νομίζω είναι κατανοητό πως για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από μικρές ε, επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις. Ε, παρόμοιες είναι καταστάσεις και στην Αυστρία. για τις μικρές αυτές επιχειρήσεις που χρειάζονται το όχημα για να πάνε στη δουλειά τους. Πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν τις εξαιρέσεις. Ε, και το ίδιο ισχύει βεβαίως και με την ε, ε, συγκοινωνία με τα εργοτάξια. Και εκεί πέρα είναι μικρές επιχειρήσεις με ένα-δύο φορτηγά που λειτουργούν σε μικρή ακτίνα. Οπότε εκεί πέρα είναι λογικό να γίνει κάτι για αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών. Μια εξαίρεση δηλαδή για να φτάσει ο κύκλος αυτός ε, ε, στα 150 ίσως και 200 χιλιόμετρα. Το δεύτερο αναφέρεται στην ε, τροπολογία 44 αυτό το οποίο πρότεινε εδώ πέρα νομίζω είναι ξεκάθαρο λέει πως θα πρέπει να υπάρξει ένα σημαδάκι για το πότε ξεκινάει η μέρα εργασίας. Και νομίζω πως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε τις απλούστερες εδώ πέρα διατάξεις της Κομισιόν. Για μένα επαρκούν και είναι ξεκάθαρες και κατανοητές κατόπιν για την τροπολογία 57. Εδώ πέρα υποστηρίζω ξεκάθαρα αυτό το οποίο αναφέρεται. Δεν επαρκεί ε, να οδηγεί σε πιθανές ποινές ο τεχνικός έλεγχος. Πρέπει να υπάρξει επιπλέον έλεγχος πριν ε, επιβληθεί ε, ποινή, δηλαδή να υπάρξει και φυσικός έλεγχος πριν πέσει το πρόστιμο. Και τελευταίο κάτι το οποίο αναφέρεται στην 89 τροπολογία εδώ πέρα λέει η Κομισιόν πως θα πρέπει ο χρόνος ε, που δεν οδηγείται να περιγράφεται ως χρόνος ε, ξεκούρασης ε, ή διαλύματος και μιλάτε εσείς εδώ πέρα για χρόνο ετοιμότητας. Εδώ πέρα θέλω μια διευκρίνηση. Τι, γιατί, τι είπα να πει χρόνος ετοιμότητας. Α, γιατί επιλέγετε αυτή την συντομηση όταν η Κομισιόν μιλάει για χρόνο ξεκούρασης και διαλύματος και είναι κάτι το οποίο είναι τελείως κατανοητό και δεν προσφέρεται για παρεξηγήσεις. Ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε εδώ πέρα γιατί έχετε αλλάξει τον όρο και συντομεύσει την διατύπωση αυτή. Ευχαριστώ. Σε Βαντάλεν. Φαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεση για την αλλαγή του κανονισμού. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Ε, αυτό για το οποίο λέτε η Κομισιόν λέει να ενσωματωθεί το σύστημα στην, στο δίπλωμα οδήγηση για να καταπολεμηθεί η απάτη και να ξέρουμε τι κάνει ο οδηγός αλλά ε, είναι υπερβολικό και δυσανάλογο το μέτρο αυτό. Γιατί μπαίνουμε και στην ιδιωτική ζωή μετά του οδηγού, όχι μόνο στο, στην επαγγελματική του. Ξέρουμε μετά πότε χρησιμοποιεί και πότε όχι, το, πότε δουλεύει και πότε όχι κτλ. Και θα ήθελα ε, να μου πει η Κομισιόν πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε κάτι τέτοιο. Ένα άλλο θέμα βέβαια σχετίζεται με τον κανονισμό, κάτι το οποίο σημαίνει πως οι πολιτικές αλλαγές ε, τις οποίες μπορούμε να ζητήσουμε είναι πολύ περιορισμένες. Το κείμενο αλλάζει, δεν μπορούμε να προσθέσουμε αυτά τα οποία θα θέλαμε ως πολιτική γιατί έχουμε απλά μία αλλαγή ε, του κανονισμού στα παραρτήματα. Η συγκήτρια. Μιλάει επίσης για την εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά εγώ νομίζω πως το θέμα εδώ πέρα αφορά περισσότερο την Κομισιόν. Η Κομισιόν μας υποσχέθηκε να μας πει τι γίνεται με την εφαρμογή για να έχουμε μια πιο εναρμονισμένη ε, εναρμόνιση. Θυμάμαι την ε, συνεδρίαση που είχε γίνει για αυτό το θέμα και μας υποσχέθηκε υψηλό βαθμός αξιωματούχος της Κομισιόν πως θα ασχοληθεί με την εναρμόνιση της εφαρμογής. Θέλω η Κομισιό να κάνει αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Εντάξει, καλή και η εκπαίδευση, οι συσκευές και τα λοιπά, αλλά όταν δηλώνουν οι αρμόδιοι για τον έλεγχο πως είναι τόσο πολύπλοκος ο κανονισμός που δεν καταλαβαίνουν πως πρέπει να λειτουργήσει, τότε κάτι δεν πάει καλά. Οπότε απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν να κάνει αυτό το οποίο είπε. Δεν θα υποβάλω ε, τροπολογίες γιατί όπως σας είπα δεν θεωρώ πως είναι στη σε η οποία ακολουθήθηκε. Η κυρία Ντιογόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αντιδράσω σε σχέση με αυτά που άκουσα για τις εξαιρέσεις. Νομίζω ότι τα προτινόμενα μέτρα δεν είναι οικονομικά μέτρα, ούτε είναι μέτρα τα οποία επηρεάζουν την προσωπική ζωή. Είναι μέτρα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Και οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του δρόμου, των δρόμων, αλλά προφανώς και των οδηγών. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους οδηγούς αυτούς από τις εξαντλητικές αυτές συνθήκες που μπορούν να μειώσουν το επίπεδο συγκέντρωσης και που μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να τους οδηγήσουν σε ατύχημα, από το οποίο ατύχημα θα είναι βέβαια αυτή τα βασικά θύματα. Ξέρετε ότι σε σύγκρουση με φορτηγό είναι ο οδηγός αυτός ο οποίος χάνει τη ζωή του πρώτος. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε εξαιρέσει. αν είναι όμως να έχουμε εξαιρέσει, αυτές θα πρέπει να γίνονται με βάση το βασικό κριτήριο της ασφάλειας και μόνο με αυτό. Και όταν άκουσα να γίνεται αναφορά σε όλους αυτούς τους άλλους επαγγελματικούς τομείς για τους οποίους θα πρέπει να γίνει μια εξαίρεση, ουσιαστικά αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδεχομένω να είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένοι οδηγώντας ένα φορτηγό αφού έχουν εργαστεί όλη την ημέρα κάπου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει η βασικό μας μέλημα να είναι η οδική ασφάλεια και ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες ευθύνες και υποχρεώσεις όχι μόνο για το αφεντικό αλλά για αυτόν ουσιαστικά που δίνει τις βασικές εντολές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, είναι τα άτομα αυτά ουσιαστικά τα οποία ε, δίνουν τις απαραίτητες εντολές προκειμένου ο οδηγός να οδηγήσει γρήγορα, να ξεπεράσει ακόμα και την προβλεπόμενη περίοδο οδήγησης προκειμένου να παραδώσει ένα προϊόν ακόμα πιο γρήγορα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα των εξαιρέσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσει με βασικότατο κριτήριο και μέλημα την οδική ασφάλεια. Και δεν θα πρέπει το κριτήριό μα να είναι εν γέννη η ε, προστασία των ρεστεχνών οδηγών. Νομίζω ότι ε, και αυτοί πάντως, λόγω της ε, επαγγελματικής κούρασης, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο και τη δική τους τη ζωή, αλλά και τη ζωή των άλλων. Νομίζω ότι το βασικό κριτήριο πάντως για τις εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Γεια σας όμως την ε, έκθεση της συναδέλφου. Θέλω να αφαιρθώ σε τρία σημεία που ε, αναφέρθηκαν. Που τα είχα αναφέρει όταν είχαμε και τη μικρή ε, κρόαση. Τώρα για την ε, άδεια οδήγησης και την ενσωμάτωσή της. Πρέπει να σκεφτούμε τις διοικητικές συνέπειες ε, για το Βέλγιο, του χάρη, αυτό σημαίνει κόστος 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν το δούμε πανευρωπαϊκά, θεωρώ πως η εκτίμηση της Κομισιόν για το διοικητικό κόστος ε, είναι πάρα πολύ χαμηλή και πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε και τι θα γίνει και, και μετά, γιατί είναι άλλο ε, το να αποσύρει κανεί μια άδεια κυκλοφορία. Αλλά αν πάρει μαζί και το δίπλωμα, τι γίνεται. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα επαγγελματικό πρόβλημα ενό ανθρώπου, ε, τιμωρείται και προσωπικά ε, και δεν έχει μετά το δίπλωμά του. Ε, θα ήθελα να αναλυθεί αυτό το, το θέμα. Δεύτερον, για τις εξαιρέσεις. να γίνουν πιο σαφείς οι εξαιρέσεις για να έχουμε και μικρότερο περιθώριο λοιπόν, γιατί οι ερμηνείες από χώρα σε χώρα είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Κοίταξε, εγώ μένω και σε μεθοριακή περιοχή. Σε μένα ε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κυπουρός ας πούμε και μεταφέρει ε, δεντράκια μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν περάσει τα σύνορα με τη Γερμανία πρέπει να έχει ταχογράφο. Αν πάει στην Ολλανδία δεν ξέρω. Νομίζω πως είναι παρόμοια η κατάσταση με το, με το Βέλγιο. Ε, οπότε πρέπει να περιορίσουμε λίγο το περιθώριο ερμηνείας ε, και για ε, αυτό το ζήτημα. Ειδικά αν μιλάμε για μια χώρα για την, όπως η Αυστρία έχουμε και συμφέρον γιατί καταλαβαίνετε αν κάνουμε την ακτίνα 100 χιλιόμετρα βγαίνουμε αμέσως εκτός συνόρων, σε όλες τις, ε, τις περιπτώσεις, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν πάει κανείς. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διασυνοριακές ε, πτυχές. Τέλος, να εκφράσω τις ε, αμφιβολίες μου όταν μιλάμε για τεχνολογία και νομοθεσία. Ήδη έχουμε τριπλές, τριπλό σύστημα συσκευών ελέγχου. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται ο έλεγχος, ποιος κάνει τον έλεγχο με κάθε σεβασμό για τους ε, αστυνομικού. Ε, γιατί τι γίνεται, πηγαίνουν οι άνθρωποι με το βιβλιαράκι για να κάνουν ερμηνεία επιτόπου των κανονισμού. Να μην καταλήξουμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου αύριο θα έχουμε πάλι μια άλλη τεχνολογία και θα έχουμε και τις τρεις υπάρχουσες. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, να υπάρξει μια συμβατότητα, όπως λέγεται, διαλειτουργικότητα και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες αναβάθμισης και να πούμε πως ε, στην τάδη ημερομηνία ε, θα πρέπει να προσαρμοστούν και όσοι δεν έχουν, αλλά 90% θα πρέπει να έχουν αυτή την τεχνολογία για να μπορεί να ελέγχεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αναρμονίσουμε τις ποινές, αλλά νομίζω μπορεί να γίνει εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου. Αυτό θα ήθελα να πω και έκανα έτσι αμέσως και τα σχόλιά μου προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Euh, Ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, thank you, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και συνέβαλαν πάρα πολύ στη συζήτηση να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για το ιδιαίτερο ανοιχτό πνεύμα που έδειξε, γιατί ήταν σε θέση να συζητήσει και να συνεργαστεί μαζί μας, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή της, καθώς επίσης και από τους συναδέλφους της. Υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποια ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε, και θα συνεχίσουμε προφανώς τη συζήτηση και με την εισηγήτρια για αυτά. Λοιπόν, κάποια συγκεκριμένα σημεία. Νομίζω ότι ορισμένοι αναφερθήκατε στο ρόλο αυτής της συσκευής. Ο βασικός ρόλος είναι να ελέγχει ότι η κοινωνική νομοθεσία εφαρμόζεται. Ζούμε όμως σε διαφορετική εποχή από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι τότε γίνανε και οι πρώτες ε, συζητήσεις. Τότε είχα πιο σκούρα μαλλιά όταν εργαζόμουν για το ζήτημα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνάδελφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν πει ότι ε, θα είχαν αντιτάξει κάποιες ε, αμφιβολίες γι' αυτό. Και τους λέω για άλλη μια φορά ότι στόχος είναι να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο μέσω της συσκευής αυτής. Εξελίσσεται όμως τεχνολογία και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία που μας δίνει αυτού του είδους η συσκευή, η οποία αρχικά είχε προβλεφθεί για τον έλεγχο του ωραρίου της περίοδου εργασίας και τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς. Το πιο σημαντικό τώρα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της συσκευή αυτής, καθώς επίσης και μια υπηρεσία γεωγραφικού εντοπισμού. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ θετικά και από μικρές επιχειρήσεις και για να καλυφθούν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε να ελέγξουμε και βλέπουμε ότι η συγγήτρια προσπαθεί να συνδυάσει τη συσκευή αυτή με τα ευφυή e συστήματα μεταφορών. Νομίζω λοιπόν ότι με τη νέα αυτή τεχνολογία που έχουμε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη νέα ευκαιρία η οποία μας δίνεται. Κάποια συγκεκριμένα τώρα σημεία. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι οι 24 μήνες είναι μια καλύτερη περίοδος από αυτή που αρχικά προβλεπόταν, προκειμένου να εισαχθεί ο ταχογράφος. Θεωρούμε ότι η πράξη καταξιοδότηση είναι ο κατάλληλος τρόπος εφαρμογής. Νομίζω ότι θέλουμε μια πιο ευθυγραμμισμένη κατάρτιση των αστυνομικών αξιωματικών ελέγχου. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλύτερους ομοιόμορφους ελέγχους κοινός ορισμός των πολύ σημαντικών παραβιάσεων. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει εδώ πέρα να προχωρήσουμε πάρα πολύ μακριά. Έχουμε και την εμπειρία από την επιβολή της νομοθεσίας. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, δηλαδή να ξεφύγουμε από τις τεχνικές, από τους τεχνικούς αυτούς ορισμούς που έχουμε και να περάσουμε περισσότερο στην νομική πτυχή του ζητήματος, όπου εκεί τίθεται και το ζήτημα ή θα πρέπει να ανοίξουμε το ζήτημα της νομικής βάσης. Ας δούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο ορισμός του σοβαρού παραπτώματος, της σοβαρής παραβίασης και στη συνέχεια να πρόκειται στα κράτη-μέλη να καθορίσουν τις κυρώσεις. Και η επεξεργασία των δεδομένων επίσης είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Πολλοί ομιλητές και η αναφερθήκατε στον συνδυασμό της κάρτας οδηγού με την άδεια οδήγηση. Ας μην συγχαίουμε όμως την προσωπική ιδιωτική ζωή με την επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου. Ας μην καταλήξουμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου θα χάσει κανείς την ευφύ αυτή κάρτα που χρησιμοποιεί επεγγελματικά και συνέχεια δεν θα είναι σε θέση καν να οδηγεί στο αυτοκίνητό του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε εμεί να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία προκειμένου να μην γίνει σύγχυση ανάμεσα στι δύο αυτέ λειτουργίε. Εναπόκειται σε εμά να βρούμε τον καλύτερο τρόπο συνδυασμού των λειτουργιών αυτών. θα πρέπει μια τέτοια διασύνδεση να μην επηρεάσει τελικά άλλες προσωπικές δραστηριότητε του ενδιαφερομένου τώρα, εξαιρέσει. Κάνοντας την πρόταση αυτή, είχαμε κατά νου και τις ιδέες που εξέφρασε η κυρία Ντουράν. Δεν λέμε εδώ πέρα ότι α, ακόμα και όταν ζει κάποιος μια δασική περιοχή θα οδηγήσει τέσσερις ώρες, θα πάει στη δουλειά του και συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψει πάλι οδήγηση τέσσερις ώρες μέχρι να πάει στο σπίτι του και ότι στην επιστροφή θα, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 30-40% θα γίνει ένα τύχημα τα, η, ιδέα των 100 χιλιόμετρων ήταν απόρρια μιας κάποιας ανάλυσης και μελέτης που κάναμε. Και ουσιαστικά προτείναμε την επέκταση αυτή για να βελτιώσουμε, να ευνοήσουμε κάποιες επαγγελματικέ δραστηριότητες. Το να προχωρήσουμε περαιτέρω από τα 100 χιλιόμετρα τώρα, ναι, μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα οδηγήσει ένα αυτοκινητόδρομο με 70 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Δεν θα πρέπει εδώ πέρα μέσω τη νομοθεσία να προκαλέσουμε προβλήματα σε όσου πρέπει να κάνουν τέτοιες, που έχουν τέτοιε επαγγελματικέ δραστηριότητε. Τώρα, όσον αφορά του επαγγελματίε αυτού οι οποίοι πρέπει να οδηγήσουν ε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή για μεγάλες αποστάσεις για να πάνε να κάνουν τη δουλειά του, να προσπαθήσαμε και, αυτό, αυτούς να τους καλύψουμε. Και γι' αυτό το λόγο θέσαμε το όριο των 100 χιλιόμετρων, λαμβάνοντας υπόψη μια περίοδο εργασίας 8 ε, ωρών και λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή στο σπίτι τους. Θα ήθελα να αφαιρθώ και σε κάποια άλλα σημεία. Έχετε λοιπόν τώρα την ε, ανακοίνωση αυτή όσον αφορά τον ταχογράφο, που είχε ως στόχο να διευκολύνει και τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους. Ας μην αγνοήσουμε την δυνατότητα μας δίνεται εδώ πέρα θα ήταν πολύ καλύτερο να μπορούμε να κάνουμε αυτόματα τους ελέγχους μέσω των συσκευών αυτών και να μην αναγκαζόμαστε να σταματάμε τα φορτηγά στο δρόμο για να κάνουμε τον έλεγχο. Τέλος. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φορείς όπως η ΣΕΜ, η ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης, που θα μπορούσαν να προτείνουν διαφορετικού τρόπου για το πώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα χωρίς να περιλάβουμε όλα στον κανονισμό. Νομίζω ότι η κυρία Φώστερ αναφέρθηκε σε αυτό. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή, το, να μεταφέρουμε κάποια στοιχεία από τα παραρτήματα στο διατακτικό του κανονισμού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον. Το θα θελήσουμε να ε, αναθεωρήσουμε τον κανονισμό αυτό, να τον προσαρμόσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς αυτό. Ας μην καταλήξουμε σε ένα ιδιαίτερα διεξοδικό και πλήρες νομοθετικό κανονισμό, ο οποίος στη συνέχεια όμως είναι ιδιαίτερα δίσκαμπτος και θα είναι αδύνατον ή πάρα πολύ δύσκολο να τροποποιηθεί. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί ω προ τη μεταφορά που κάνουμε από τα παραρτήματα προς το διατακτικό του κανονισμού. Α μην προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όλα τα κοινωνικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που υπάρχουν μέσω ενός τεχνικού ουσιαστικά κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τέλος το λόγο έχει η αλλα προβληματα που υπαρχουν μεσω ενο τεχνικου ουσιαστικα κανονισμου σα ευχαριστω ευχαριστουμε πολυ και τελος το λογο εχει η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και την Επιτροπή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρόθεσή μας είναι να βελτιώσουμε τον ψηφιακό ταχογράφο έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ε, όργανο φιλικό προς το χρήστη γιατί σήμερα δυστυχώς ο ταχογράφος δεν δίνει πολλές πληροφορίες στον οδηγό. Θα θέλαμε στο μέλλον ο ταχογράφος να είναι πολύ πιο χρήσιμος και για τον οδηγό έτσι ώστε να μπορεί να τηρήσει την κοινωνική νομοθεσία. Θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ με την κυρία Ντουράν. Ο βασικός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια. Θα ήθελα να διαγραφούν οι εξαιρέσεις προσωπικά και νομίζω ότι τα 50 χιλιόμετρα ήταν το πιο σωστό όριο. Από όσο ξέρω η Επιτροπή έχει διενεργήσει μία μελέτη και τα 100 χιλιόμετρα είναι το ύψιστο όριο. Βεβαίως εδώ θα υπησέλθουν πολλές τροπολογίες και με τη λήξη των 50 ε, χιλιόμετρων γίνονται άλλες εξαιρέσεις και αυξάνουμε μέχρι τα 200 χιλιόμετρα. Ελπίζω οι συνάδελφοι να προβάλλουν άλλες προτάσεις περιοριστικές σε σχέση με τα διάφορα συνεργεία και τις επιχειρήσεις μεταφορών. Διαφέρει κατάσταση στα κράτη-μέλη. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και συνεργεία και ακόμα πολύ ενδιαφέρον την άποψη των συναδέλφων. Υπάρχουν άλλες χώρες όχι που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το πλαίσιο, αλλά υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός, ένας πλήρης διαχωρισμός μεταξύ συνεργείων και επιχειρήσεων μεταφορών. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν να υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ αυτής της ε, θέσης. Ξέρω όμως ότι θα έχουμε πολλές τροπολογίες και μαζί με τους συναδέλφους θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο διευθέτησης. Επίσης, για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων έχουμε βελτιώσει το κείμενο και να μην υπάρχουν αυτόματες κυρώσεις ως προς την ενσωμάτωση, όπως είπε και η Κομισιόν. Τη στιγμή που θα γίνει αυτή η συγχώνευση, δηλαδή της εφιούς κάρτας και της άδειας οδήγησης, αυτό δεν θα πρέπει να πλήξει τον οδηγό. Δηλαδή, εάν υπάρχει απλή κύρωση, αυτό δεν θα πρέπει να πλήξει την χρήση της άδεια οδήγηση του οδηγού ιδιωτικά. Και αυτό το λέω γιατί στο ενσωματωμένο σύστημα μηχανογράφησης όπου θα έχουν πρόσβαση και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Μεταφορών ε, το κάθε Υπουργείο θα μπορεί να σπληρώνει τα στοιχεία. Δηλαδή, μιλάμε για κυρώσεις, ότι έρεται η άδεια οδήγησης για ένα χιχρονικό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία θα ενυπάρχουν, θα εισαχθούν στο ενιαίο σύστημα και θα τη χάνουν εύκολης επαλήθευσης. Και νομίζω ότι από τεχνικής πλευράς μπορεί να γίνει αυτή η ενσωμάτωση και όπως είπε και η Κομισιόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρης ε, προετοιμασία. Θα πρέπει να γίνει μια μελέτη αντικτύπου έτσι ώστε τη στιγμή που θα γίνει η συγχώνευση να γίνει κατά σωστό τρόπο και ίσως να γίνει και βαθμιαία ε, κλιμακωτά έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη. Είναι γεγονός ότι ως προσορισμένα ερωτήματα των συνοδέλφων θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει η έννοια της ε, διαθεσιμότητας, γιατί όταν ένας οδηγός βρίσκεται στην επιχείρηση και κάνει ορισμένα γραφειοκρατικά δεν ε, αναπαύεται. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να πληγεί η έννοια της ανάπαυσης και η ώρα εργασίας. Ως προς τα παραρτήματα, Έχω λάβει μόνο ορισμένα στοιχεία των ε, παραρτημάτων που θεωρώ σημαντικά. Βεβαίω, μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων η Κομισιόν μπορούσε να αλλάξει τα παραρτήματα γενικά. Δυστυχώς υπάρχουν όμως ε, τεχνικές προδιαγραφές ύψης της σημασίας που έχουν αλλάξει δέκα φορές. Την τελευταία φορά άλλαξαν το 2009 και η Επιτροπή αναγνώρισε σε συζητήσεις ότι ορισμένα τμήματα των παρατημάτων δεν είναι επίκαιρα. Το Συμβούλιο θέλει να διαγραφούν τα παραρτήματα μέσα σε μια μεταβατική περίοδο και μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων να δούμε ποια στοιχεία πρέπει να ενταχθούν στον ίδιο τον κανονισμό για να ορίσουμε επακριβώς την εντολή των ε, κατεξουδότηση πράξεων. Θα σταματήσω εδώ, περιμένω τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων, δέχομαι οποιαδήποτε συζήτηση, υπόδειξη. Είχαμε και την ακρόασή μας και την συνάντηση με τα συνδικάτα των επαγγελματιών οδηγών και με το GRC θα ήθελα να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία ενιαία λύση για να πληροφορήσουμε και τα συνδικάτα. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τους συναδέλφους, περιμένω τις τροπολογίες σας και είμαι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσικάου. Η προθεσμία είναι η 15η Μαρτίου για τις τροπολογίες. Κυρία Φώστερ, θέλετε κάτι? Με συγχωρείτε. Έφυξα ένα θέμα που αν με ανησυχεί σε πολλά κράτη-μέλη. Για τους Ουκρανούς και Ρώσους οδηγούς που οδηγούν στην Ευρώπη. Τι θα κάνετε, γιατί όλα αυτά τα κάνουμε για τους Ευρωπαίους μεταφορείς. Τι θα κάνετε σε τέτοιες ε, καταστάσεις και περιστάσεις. Δεν μου απάντησε κανείς, ούτε η κυρία Τσικάου, ούτε η Επιτροπή. Μπορείτε να μου πείτε ή ο ένας ή ο άλλος. Ε, Θέλει κάτι να πει η Επιτροπή. Ε, πρέπει να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την Παρασκευή μάλιστα το συζητάμε στη Γενέβη, στον ΟΗΕ. Υπό το πλαίσιο του AETR ε όπως το λέμε. Ανησυχούν βεβαίως ότι τους, τους επιβάλλουμε το έξτρα κόστος του ψηφιακού ταχογράφου. Πρέπει να τους πείσουμε για το όφελος. Αλλά θα το συζητήσουμε στον ΟΗΕ, οπότε θα φροντίσουμε να εφαρμόσουν ε, τα ίδια πράγματα, να έχουν τον ίδιο εξοπλισμό που έχουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Κυρία Τσεκάου. Και στο 17, στο έχοντας υπόψη 17, κυρία Φώστερ, θέλετε να μ' ακούσετε. Υποβάλλετε ερωτήσεις, αλλά δεν ακούτε. Και στην αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού γίνεται μνήα σε αυτή την ε, συμφωνία AETR με βάση τα Ηνωμένα, Έθνη και οι, από τις όμερες χώρες οι, οι οδηγοί χρησιμοποιούν τα μηχανήματα του παραρτήματος 1β. Σας ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 15 Μαρτίου δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, άρα σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα συνεδριάσουμε στις 26 Μαρτίου στις 5